Καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλους. Ακόμα και αν δεν είμαστε πολύ άριθμοι στη συνειδρίαση αυτή, πιστεύω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, περνάμε στο πρώτο σημείο της μερισιας διάταξης, έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Σας προτείνω μία μικρή αλλαγή. Το σημείο 8, ισότητα των θύλων και ενδυνάμωση των γυναικών στην ψηφιακή εποχή, θα το εξετάσουμε μετά το σημείο 10. Δεν προτείνω άλλες τροποποιήσεις στην ημερήσια διάταξη. Πέρα από αυτήν, να συμφωνείτε λοιπόν, μπορούμε να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Περνάμε στο σημείο 2, ανακοινώσεις της Προέδρου. Στις 12.30 σήμερα, έξω από την αίθουσα αυτήν, θα γίνει μία μικρή δεξίωση από την Μονάδα Ισότητας των Θήλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μας έχουν καλέσει να συμμετάσχουμε σε αυτή τη δεξίωση. Λοιπόν, αυτά λάβει η χώρα που σας είπα εκτός αιθούσης αυτής στις 12.30. Περνάμε στο σημείο 3 της ημερήσιας διάταξης. όπου εδώ εξετάζουμε την έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2010-18 του Συμβουλίου της 8 Μαρτίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της αναθωρημένης συμφωνίας πλαισίου για τη γονική άδεια που συνήφθη από τις οργανώσεις Business Europe, UEAPME, CEP και την Ευρωπαϊκή Στομοσπονδία Συνδικάτων. Εγώ είμαι η συγγήτρια, συντάκτρια μάλλον της γνωμοδότησης αυτής Μπορώ λοιπόν εγώ να κάνω στην αρχή κάποια εισαγωγικά σχόλια και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η συζήτηση. Μα ζητήθηκε λοιπόν να συντάξουμε μία γνωμοδότηση. Η καθήλυνα αρμόδια επιτροπή είναι η Επιτροπή Απασχόληση. Προσπαθήσαμε λοιπόν να καταλήξουμε σε μία κάποια συμφωνία με του συναδέλφου από την Επιτροπή αυτή. Ξέρετε ότι εμεί είχαμε ζητήσει στην αρχή να είμαστε η καθήλυνα αρμόδια επιτροπή για την έκθεση αυτή, αλλά η Επιτροπή Απασχόληση, η διαφορετική άποψη, θεωρούσε ότι ήταν δική του αρμοδιότητα. Η συμφωνία λοιπόν στην οποία καταλήξαμε είναι εμείς να συντάξουμε απλώ μια γνωμοδότηση. Σας τα λέω τώρα όλα αυτά, διότι πολύ συχνά όταν συντάσσουμε τέτοιε γνωμοδοτήσει. ξέρετε ότι πρέπει να πληρούμε συγκεκριμένες προποθέσει. Οι γνωμοδοτήσει δεν πρέπει να είναι ιδιαίτερα εκτενεί. διότι αν είναι ιδιαίτερα μακροσκελής ε, οι γνωμοδοτήσει τότε αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι ε, πολλά από αυτά τα οποία προτείνουμε στις νομοδοτήσεις τελικά δεν συμπεριλαμβάνονται στο τελικό κείμενο της καθήλυνα αρμόδιας επιτροπής. Μολονότι λοιπόν γνωρίζω ότι υπάρχουν πολλές διαφορετικές ιδέες που θα μπορούσαμε να υποβάλουμε για το συγκεκριμένο αυτό θέμα, είναι πάρα πολύ σημαντικό να πρέπει να μπορούμε τελικά να επικεντρωθούμε στα πιο κέρια σημεία. Τα σημεία που θεωρούμε ότι αποτελούν πραγματική προτεραιότητα για την Επιτροπή μας έτσι ώστε τουλάχιστον οι προτεραιότητες αυτές να συμπεριληφθούν εν τέλει στο κείμενο της Επιτροπής ε, Απασχόλησης. Ξεκινάω καταρχάς με δύο προτάσεις όσον αφορά την ε, αιτιολογική σκέψη, όπου λέμε ότι ο στόχος της απασχόλησης 75% που τίθεται στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική 2020 έχει επιτευχθεί για τους άνδρες, αλλά είναι απίθανο επιτευχθεί ο στόχο αυτό για τι γυναίκε μέχρι το 2020. Οι γυναίκε αυτή τη στιγμή έχουν ένα ποσοστό απασχόληση τη τάξη του 63,5%. Αν δεν υπάρξουν λοιπόν μέτρα για να υποστηριχθεί η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασία, δεν πρόκειται με τίποτα να πετύχουμε μέχρι το 2020 το ποσοστό απασχόληση 75%. Επίση λέμε ότι η γονική άδεια με χαμηλέ αποδοχέ δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ιδιαιτέρω τελικά και αυτό είναι σαφές τουλάχιστον για τους πατέρες, οι οποίοι ε, όταν παίρνουν γονική άδεια, άδεια πατρότητας, ε, την παίρνουν για ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα και μόνο εφόσον ε, είναι μεταβιβάσιμες αυτές οι περίοδοι άδεια και συνήθως βέβαια μεταβιβάζουν το δικαίωμά τους αυτό στις γυναίκες τους. Επίσης, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat για το 2010, περίπου 3.500.000 γονείς έκαναν χρήση γονικής άδειας ενώ μόνο 94.800 από αυτούς ήταν άνδρες και οι γυναίκες ήταν 3.400.000 περίπου. Βλέπετε λοιπόν ότι όταν έχουμε μια γονική άδεια η οποία είναι μεταβιβάσιμη και η οποία συνοδεύεται από χαμηλές αποδοχές για την περίοδο αυτή, τελικά καταλήγουν οι γυναίκες να κάνουν χρήση της άδειας αυτής. Ζητούμε λοιπόν από τους κοινωνικούς εταίρους να αναγνωρίσουν την ε, αποτυχία της οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη γονική άδεια. Δεν έχει επιτύχει αυτή η οδηγία του στόχου της και θεωρούμε ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί, να ενεργοποιηθεί η ρήτρα αναθεώρησης για να αναθεωρηθεί η οδηγία αυτή, κυρίως με την έγκριση μέτρων τα οποία θα θεσπίζουν επαρκή και βάση κινήτρων οικονομική αποζημίωση για την απώλεια εισοδήματο, που υφίστανται οι γονεί που κάνουν χρήση γονική άδεια. Επίση, η γονική άδεια θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ω εξατομικευμένο δικαίωμα, μεμονωμένα για τι γυναίκε και του άντρε, και να μην αντιμετωπίσετε πάντα ω μια γονική άδεια η οποία είναι μεταβιβάσιμη και που τελικά περνάει πάντα από του άντρε στι γυναίκε. Αυτό είναι το αρχικό κείμενο το οποίο σας προτείνω. Θα υποβάλω επιπλέον τροπολογίες για να συμπεριλάβουμε επιπλέον στοιχεία στην όλη αυτή η συζήτηση και νομίζω ότι θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε την υφιστάμενη συγκυρία. Ενδεχομένω θα μπορούσαμε να είχαμε ακόμα και κάποιε περαιτέρω προτάσει από την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ξέρετε ότι επί του παρόντο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεξεργάζεται την οδηγία για την άδεια μητρότητα Καθώ επίση και κάποιε άλλε προτάσει οι οποίε αποσύρθηκαν σε μία πρώτη φάση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τώρα μα λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα επανέλθει με περαιτέρω πιο ενισχυμένε προτάσει για αυτά τα ζητήματα και ότι όλα αυτά θα ενταχθούν στο γενικότερο πλαίσιο τη γονική άδεια. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία αυτή που μα δίνεται, αυτή τη χρονική περίοδο, προκειμένου να στείλουμε μέσω της έκθεσης αυτής ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ένα συγκεκριμένο μήνυμα προ τα έξω. Και εμεί ω Επιτροπή Γυναικών μπορούμε να δώσουμε κάποια καθοδήγηση στην Επιτροπή Απασχόληση. Νομίζω ότι θα πρέπει να αναφερθούμε επίση στο ζήτημα τη ανισότητα ανδρών και γυναικών στην αγορά εργασία, το μισθολογικό χάσμα που υπάρχει μεταξύ ανδρών και γυναικών. Ξέρετε ότι το μισθολογικό χάσμα κατ' επέκταση οδηγεί και σε συνταξιοδοτικό χάσμα στη συνέχεια. Καταλήγουν τελικά πάντα οι γυναίκε να αυτέ οι οποίε φροντίζουν κατά κύριο λόγο τα παιδιά είναι οι γυναίκες αυτές οι οποίες χρησιμοποιούν κυρίως τα δικαιώματα γονικής άδεια, αλλά στα πλαίσια της ισότητας στην αγορά εργασίας θα έπρεπε να υπάρχει κανονικά μια καλύτερη ισορροπία ανάμεσα στη χρήση που γίνεται μεταξύ ανδρών και γυναικών όσον αφορά τη γονική άδεια. Με άλλα λόγια, τόσο οι άντρε όσο και οι γυναίκε θα έπρεπε ισότιμα να χρησιμοποιούν τα δικαιώματα γονικής άδεια. Θέλουμε λοιπόν και για τη γονική άδεια μεγαλύτερη και πιο ισχυρή ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Νομίζω λοιπόν ότι ως προς αυτό θα πρέπει να έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες θα γίνουν ακόμα πιο σαφείς όταν θα έχουμε και τις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι σημαντικό λοιπόν να ενισχυθεί η χρήση της γονικής άδεια. Ξέρω ότι τα πράγματα διαφέρουν πολύ από τη μία χώρα στην άλλη. Είναι σημαντικό να επιτρέψουμε το απαραίτητο χρονικό διάστημα για να προσαρμοστούν οι εθνικές νομοθεσίες. Πρέπει να είναι σαφές πάντως ότι θα πρέπει σύντομα να έχουμε ένα δεκαετές το πολύ πλαίσιο το οποίο θα επιτρέπει στα κράτη-μέλη να προσαρμόσουν τις εθνικές νομοθεσίες, να καταλήξουν δηλαδή σε συστήματα γονικής άδεια τα οποία θα συνοδεύονται από αξιοπρεπείς αποδοχές και τα οποία θα χρησιμοποιούνται τόσο από τις γυναίκες όσο και από τους άντρες. Αυτά είχα να πω στην εισαγωγική μου αυτή παρέμβαση. Μπορούμε να ξεκινήσουμε τώρα τη συζήτηση. Θα ήθελα να δω και ποια είναι η δική σας άποψη. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσίαση που κάνατε. Χαίρομαι πάρα πολύ που μπορώ να συμμετάσχω στη συζήτηση ως μέλος και της Επιτροπής Απασχόλησης αλλά και της Επιτροπής Γυναικών. Βλέπουμε εδώ ότι οι γυναίκες βουλευτές υποστηρίζουν αυτή τη θέση για τη γονική άδεια να είναι μεταβιβάσιμη διότι ο στόχος μας είναι να υποστηρίξουμε το σύνολο της οικογένειας. Θέλω να τονίσω πόσο σημαντικό είναι αυτό και θα το εκφράσω και στις ε, τροπολογίες μου. Γιατί ο στόχος ε, εν τέλει της γονικής άδειας είναι να φροντίζει ε, ένας από τους γονείς το παιδί. Η παράταση της άδειας από τέσσερις σε έξι μήνες έχω την εντύπωση ότι ίσως δεν είναι αυτό που αρμόζει να προτείνουμε. Νομίζω ότι θα ήταν προσφορότερο να έχουν περιθώριο ελιγμών τα κράτη-μέλη και να διαμορφωθεί το σύστημα σε εθνικό επίπεδο σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους. Σε σχέση με τη μη μεταβασιμότητα αυτής της παράτασης ή Ολόκληρη τη διάρκεια είναι λεπτό ζήτημα για μένα. Νομίζω ότι οι γονεί οι ίδιοι θα πρέπει να έχουν τη διακριτική ευχαίρεια να αποφασίσουν. Θα ήθελα επίσης να τονίσω πως πρόκειται εδώ για ένα κανονισμό πλαίσιο Δεν εκδίδουμε εδώ κατευθυντήριες γραμμές, προσπαθούμε να διαμορφώσουμε ένα πλαίσιο Στη συνέχεια θα δούμε πώς θα εφαρμοστεί αυτό σε επίπεδο κράτους μέλους. Σε κάθε περίπτωση επιδέχεται βελτίωση η πρόταση. Χρειαζόμαστε καλύτερους, ευνοϊκότερους όρους για τη χρήση της γονικής άδειας, για την επιστροφή τους στην αγορά εργασίας. Ε, αυτά υποστηρίζει το ΕΛΚ και Προς αυτή την κατεύθυνση θα καταθέσουμε και τροπολογία. Σας ευχαριστούμε και πάλι για την παρουσίασή σας. Σας ευχαριστώ. Κυρία Σούπερ. Ευχαριστώ. Εν γέννη συμφωνούμε με την πρόταση έκθεσης, το σχέδιο έκθεσης. Ε, αποδίδεται ιδιαίτερο ειδικό βάρος και δικαίως στο θέμα των πληρωμών. Δεν μπορούμε να αποφύγουμε αυτό το βασικό σημείο, δηλαδή καταβολή κατά 100% του μισθού κατά τη διάρκεια της γονικής άδειας ή σε ένα ποσοστό ε, που πλησιάζει το 100%. Χρειάζεται αυτή η ειδική άδεια για να μπορέσουν όλοι να συνεχίσουν τη ζωή τους ε, ενώ ταυτόχρονα αυξάνονται οι δαπάνες με την έλευση του παιδιού. Τέτοια, τέτοιοι μηχανισμοί υπάρχουν σε διάφορες χώρες. Σε άλλες όχι και αυτό πραγματικά είναι άδικο. Γι' αυτό θα θέλαμε να αναθεωρηθεί η οδηγία για να δοθεί η απαιτούμενη έμφαση στο θέμα των πληρωμών. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε και τη θέση των κοινωνικών εταίρων. Η μεγάλη τους πλειοψηφία τάσσονται υπέρ της θέσης αυτής. Κάτι άλλο. Σε χώρες όπως η Πορτογαλία γνωρίζουμε πολλές περιπτώσεις ε, ε, γονιών που ε, λαμβάνουν αυτή τη γονική αδεία, κυρίως πρόκειται για τον πατέρα, παίρνουν την πατρική άδεια και ε, παρόλα αυτά συνεχίζουν να εργάζονται για να έχουν ε, καλύτερε συνθήκε για να μεγαλώσουν τα παιδιά. Ε, αυτό σχετίζεται με το μισθό και σχετίζεται με το πρόβλημα των πληρωμών που προανέφερα. Θέλουμε λοιπόν να συμπεριληφθεί και αυτό το στοιχείο, τα στοιχεία που έχουμε δηλαδή για τέτοια φαινόμενα. Για τον οδικό χάρτη τώρα ε, που μας προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποσύρει ε, την άδεια για τη μητρική άδεια και αυτό ε, εγκυμονεί κινδύνους. Δεν λέει τίποτα αυτό ο ειδικός χάρτης. Ε, είναι ένα ευχολόγιο. Προθέσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι πρέπει να είναι αναλογικά και αποτελεσματικά τα μέτρα, Χωρί όμω να εξασφαλίζεται η επιτυχία των μέτρων για την αγορά εργασία παραδείγματος χάρη, να έχουμε πιο ευέλικτε μορφές εργασίας. για να μπορέσει να υπάρξει βέλτιστη δυνατή χρήση της ε, γονικής άδειας. Θα έπρεπε λοιπόν να καταθέσουμε εμείς προτάσεις ε, συμπληρώνοντας ε, τον οδικό χάρτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να κατοχυρώσουμε αυτά τα δικαιώματα. Κάτι άλλο. Μας λέει η συγγήτρια ότι πρέπει να υπάρξει ισότιμη κατανομή των μη μεταβιβάσιμων ε, τμήματων της γονικής άδειας. η η ίσω ίσως θα έπρεπε να καταθέσει μια συγκεκριμένη πρόταση για την ε, ισότιμη κατανομή του χρόνου, για την ε, μη μετεβάσιμη άδεια. Ε, υπάρχουν χώρες όπου είναι ιδιαίτερα αυστηρές οι λύσεις ε, και είναι πολύ περίπλοκοι μηχανισμοί, το πλαίσιο, οι διατάξεις που ισχύουν, οπότε ε, θα πρέπει να έχουμε μια υποχρεωτική διάρκεια των μη μεταβάσιμων τμήματων της άδεια. Συμφωνώ λοιπόν για να γίνει η σύσταση για την ισότιμη κατανομή, αλλά δεν ξέρω αν πρέπει να υπάρχει ε, μια υποχρεωτική διάρκεια για το μη μεταβάσιμο κομμάτι. Υπάρχει ελάχιστη διάρκεια ε, το τετράμινο επίσης. Και μιλάμε για την παράταση κατά δύο μήνες. 20 εβδομάδες μητρική άδεια και 4 πατρική. Και η συνολική περίοδος θα είναι 6 ε, μήνες και ε, κατόπιν κάθε κράτος μέλος ε, μπορεί να αποφασίσει με ποιο τρόπο θα εφαρμόσει αυτό το σύστημα. Δεν έχω καταλάβει ακριβώς πώς θα γίνει αυτό. Μου δημιουργήθηκαν αμφιβολίες ακούγοντάς σας, αν κάνετε την παρουσίαση. Σας ευχαριστούμε. Η κυρία Βάρνα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την καταπληκτική της παρουσίαση για μας, τους πρασίνους. Είναι ξεκάθαρη η θέση μας, είναι πολύ καλή η βάση για τις πελλοντικές εργασίες. Πρέπει να συμφιλιώσουμε την οικογενειακή και την επαγγελματική ζωή για τους άντρες και για τις γυναίκες. για την ε, ε, ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας αλλά και για την καταβολή των πληρωμών ε, για την αμοιβή της μη αμοιβόμενη εργασίας στο σπίτι γιατί είναι θέμα ίσης μεταχείρισης και ίσης θέσης της γυναίκας στην αγορά εργασίας. Λέτε στην παρουσίασή σας ότι υπάρχουν και τα συμπεράσματα ε, της αξιολόγησης και ότι είναι αποθαρρυντικά τα αποτελέσματα και ε, ε, ξέρουμε όλοι ότι δεν υπάρχει ακόμη η δέουσα συμφιλίωση της οικογενειακής και της επαγγελματική ζωής και δεν εφαρμόζουν σωστά οι ποσοστός, δεν ενσωματώνονται σωστά οι γυναίκες στην αγορά εργασίας και μαθαίνουμε ότι υπάρχουν στατιστικά στοιχεία που δείχνουν ότι δεν ότι βελτιώνονται οι ποσοστώσεις των γυναικών, αλλά ε, νομίζω ότι είναι πολύ κοινικό αυτό. Τι σημαίνει ε, ότι ε, έχουν υψηλότερα τελικά ποσοστά ανεργίας οι οι γυναίκες έχουν ε, μεγαλύτερα ποσοστά μερικής απασχόλησης. Ενώ φαίνεται δηλαδή στις στατιστικές ότι βελτιώνεται η θέση τους, ουσιαστικά δεν ισχύει αυτό, δεν είναι θετική η τάση, διότι ε, δεν επιτυχάνεται έτσι η πλήρης ενσωμάτωσή του στην αγορά εργασίας, ε, διότι δεν είναι ικανοποιητικές οι θέσεις εργασίας που έχουν. Στη συνέχεια, διαπιστώνουμε ότι απομακρύνονται οι γυναίκες από την αγορά εργασίας για να φροντίσουν τα παιδιά και πρέπει να εξασφαλίσουμε την επιστροφή τους με μια κατάλληλη αμοιβή μετά το πέρας της άδεια. Όλα αυτά που τονίσατε μέσα στην έκθεσή σας τα υποστηρίζουμε, ζητάτε αναθεώρηση της οδηγίας. Νομίζω ότι έχουμε μία σειρά άριστων μέτρων προτείνεται, ε, όπως παραδείγματο χάρη ε, η παράταση της διάρκειας από τις 4 6 εβδομάδες ε, και η αντιστάθμιση ως προς την αμοιβή, ως προς το μισθό έχουμε ε, παρατηρήσει ότι όσο αυξάνονται οι δυνατότητες ε, για τα ε, κέντρα φροντίδας των παιδιών, για τους παιδικούς σταθμούς, για την μητρική άδεια, τόσο περισσότερο αυξάνεται και η γενετικότητα. Αποφασίζουν οι γυναίκες να κάνουν παιδιά. Ε, στις 14 ε, Δεκεμβρίου θα έρθει η κυρία Γιώργα στην, στο Κοινοβούλιο για να συζητήσουμε αυτό το ζήτημα. Θα πρέπει λοιπόν να ε, δράξουμε αυτή την ευκαιρία και να ε, στρεφόμενοι προς το μέλλον να συζητήσουμε αυτό το τόσο σημαντικό ζήτημα. Ευχαριστώ. Αυτά που ακούσαμε συνδέονται και με τη δική μου έκθεση, αλλά διαρωτώ με, μπορούμε να πούμε δύο λόγια για τι συζητήσει σα με, τη, με τα συνδικάτα και τη θέση των συνδικάτων για το θέμα. Να μας πούν τι προκλήσεις ε, αντιμετωπίζουν. Για να δούμε δηλαδή αν προωθούνται έτσι και άλλα συνδικαλιστικά θέματα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κυρία Πρόεδρε, ως εισηγήτρια πιστεύω ότι θέσατε σαφέστερα τις προτεραιότητες. Πρώτον, η αμοιβή, όταν μιλούμε για συγκερασμό επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, και το θέμα των νομανικών αδειών, ε, εννοείται ότι το θέμα της αμοιβή έχει να κάνει με την φτώχεια. Γιατί την φτώχεια των γυναικών Δείτε οι γυναίκες ε, δεν πληρώνονται για τον ε, χρόνο κατά τον οποίο δεν δουλεύουν με την τεχνική έννοια του όρου. Σήμερα έχουμε εταιρείε οι οποίε δεν εξασφαλίζουν καμία ισορροπία γιατί ε, εν τέλει αυτοί οι οποίοι βγαίνουν χαμένοι επίσης είναι και οι άντρες. Μπορούμε να μιλήσουμε εδώ στην Επιτροπή Γυναικών για το θέμα. Είναι μια προβληματική που αφορά γενικότερα την κατανομή του χρόνου εργασία μεταξύ προσωπική και επαγγελματική ζωή. Λοιπόν, ένα γενικότερο θέμα. Γύρω φαν έχει κάνει μια μελέτη και στην οποία περιγράφουν αυτά τα οποία αντιμετωπίζουν οι άντρες και στην δουλειά. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια συνοχή μεταξύ των ε, αδειών. Σύμφωνα με την μελέτη, οι τρεις προσεγγίσεις, μητρική, πατρική, γονική άδεια, δεν αποτελούν ένα συνεκτικό σύνολο. Σήμερα όλα αυτά δείχνουν ότι η λήψη της γονικής άδειας αφορά κατά κύριο λόγο τις γυναίκες παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει στον τομέα. Αυτές οι τρεις λοιπόν προτεραιότητες είναι σημαντικές. Επίσης στην έκθεση λέτε για τις νέες μορφές οικογένειας. Περί πρόκειται, έχουμε χωρισμένες, χωρισμένες ζευγάρια, τα οποία το θέμα περιπλέκεται, το πώς κατανέμεται δηλαδή η γονεϊκή άδεια. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να λάβουμε επίση υπόψη μας. Α μην ξεχνούμε ότι στι μέρες μας μία στι τρεις οικογένειε ζει χωριστά. Οπότε πρέπει να λάβουμε υπόψη μας αυτή τη νέα πραγματικότητα όταν μιλάμε για γονεϊκή άδεια. Κυρία Νόλτ, έχει τον λόγο. Θέλω να πω κάτι σχέση με την ορολογία, τη γλώσσα που χρησιμοποιούμε εν προκειμένου. Μιλούμε για γονική άδεια. Μήπως ο όρος αυτός δεν είναι ο καλύτερος. Μιλούμε για χρόνο, όχι για άδεια. Πρόκειται για χρόνο στην πραγματικότητα και δεν ξέρω στις άλλες χώρες τι γίνεται. Χρησιμοποιείται όρος άδεια ή όρος χρόνος. Βέβαια, για το οικογένειο ο χρόνος αυτός φαίνεται ως άδεια, αλλά δεν πρόκειται, περί αυτού πρόκειται για χρόνο για τους γονείς. Πρόεδρος, τι να σου πω, τώρα από ότι για άδεια διακοπές, ε, δεν ξέρω, δεν, δεν ξέρω για ποιον όρο λέτε, γιατί υπάρχουν διάφορες μεταφράσεις αλλά σίγουρα θα το προσέξουμε το θέμα. Λοιπόν, να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους και τις συναδέλφους για τις παρεμβάσεις τους. Εν γέννη, νομίζω, συμφωνούμε περί του ποιοι είναι οι κύριοι στόχοι. Είμαστε τυχεροί πάντως στην Επιτροπή αυτή, διότι από ό,τι διαπιστώνω τουλάχιστον έχουμε την κυρία Αρένα, η οποία είναι αρμοδία για το θέμα στην Επιτροπή Απασχόληση, στην ΕΜΠΛ, την καθήλυνα αρμοδία επιτροπή, η οποία θα μα βοηθήσει. Γιατί πολλά από τα στοιχεία που καταθέτουμε εδώ θα ενσωματωθούν στο κείμενο τη έκθεση. Δύο ακόμη θέματα. Σε απάντηση κάποιων σχολείων. Είναι αλήθεια ότι αυτή τη στιγμή και τεκμηριώνεται αυτό και από τα στοιχεία τα αριθμητικά στην έκθεση, ότι δίνουμε ακόμη μάχη για δικαιώματα τα οποία πρέπει να είναι μεταβιβάσιμα. Δεν ξέρουμε ποια διατύπωση θα το υποστηρίξουμε αυτό, αλλά γενικά για τον στόχο συμφωνούμε. Να εξηγήσω γιατί χρειάζεται περισσότερη δουλειά εδώ. Στην Ισπανία δεν υπήρχε προσωπική μη μεταβιβάσιμη άδεια στην Ισπανία. Στην πραγματικότητα μόνο 2% των ε, πατεράδων έκανα χρήση αυτή τη δυνατότητα. Μόνο 2%. Γιατί είναι καθιερωμένη η ιδέα, το στερεότυπο, ότι τελικώ την άδεια πρέπει να την παίρνουν οι γυναίκε και ότι αυτό δεν είναι δουλειά των ανδρών. Εν τούτης, όταν θεσπίστηκε η σχετική νομοθετική τροποποίηση, όταν δόθηκαν δύο εβδομάδε μόνο για τον πατέρα, με πλήρη αμοιβή, μη μεταβιβάσιμη, τότε 80% των ε, πατεράδων πήραν τη σχετική άδεια. Το ότι έκαναν χρήση λοιπόν δείχνει ακριβώς ότι μέσω της νομοθεσία μπορούμε να φέρουμε πιο κοντά τα δικαιώματα ανδρών και γυναικών μέσω μη μεταβιβάσιμων ακριβώς δικαιωμάτων. Αυτό σημαίνει περισσότερη ισότητα και στην ανατροφή των παιδιών, αλλά και στην αγορά εργασίας εν γέννη. Ξέρω ότι είναι λεπτό το ζήτημα, αλλά πρέπει να πάμε παρακάτω. Πρέπει να αλλάξουμε. Γι' αυτό, όπως προείπα, χρειάζεται ένα ευέλικτο χρονοδιάγραμμα, διαφορετικό ενδεχομένω σε κάθε χώρα για να αξιοποιήσουμε αυτήν την ευκαιρία ώστε σύν χρόνο να προσφέρουμε περισσότερη ισότητα όταν πρόκειται για αγωνικέ άδειε. Δεν λέω ότι χρειάζεται περισσότερο χρόνο, περισσότερη άδεια, δεν λέω ότι πρέπει να είναι περισσότερο ή λιγότερο. Αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Ούτω ή άλλω σε κάθε χώρα έχει θεσπιστεί αριθμό εβδομάδων γονική άδεια. Από εκεί πέρα το θέμα είναι ευελιξία με στόχο περισσότερη ισότητα σε όλους τους τομείς. Αυτή είναι η κεντρική ιδέα. Αυτό πρέπει να είναι και το μήνυμά μας, το χειρό μας μήνυμα. Ας προσπαθήσουμε να τα ενσωματώσουμε όλα αυτά στο κείμενο για να τα στείλουμε στην Αρμόδια Επιτροπή. Είμαι εδώ, διαθέσιμη η συζήτηση, ώστε να πετύχουμε, όπως είπα, την καλύτερη δυνατή διατύπωση. Τώρα, όσον αφορά τη σημερινή Σήμερα εξετάσαμε το σχέδιο προθεσμία για το 11 Ιανουαρίου, ψηφορία στην Επιτροπή στις 17 Φεβρουαρίου. Ψηφορία στην Επιτροπή 17 Φεβρουαρίου. Επόμενο σημείο στη ημερήσια διάταξη. Το οποίο είναι η έκθεση επίτευξη του στόχου της φτώχειας Στάκτρια γνωμοδότησης η Julie Ward πρόκειται για νομοδότηση επαναλαμβάνω για έκθεση της Επιτροπής ΕΜΠΛ κύριε Ward αυτό το λόγο Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε Είμαι πραγματικά ευγνώμων που μου δόθηκε η δυνατότητα να ασχοληθώ με το πολύ σημαντικό αυτό θέμα, ιδίω στην τρέχουσα αυτή περίσταση, καθότι αναθεωρείται τώρα η Ευρωπαϊκή Στρατηγική 2020. Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν δώσει νέα πολιτική όθηση για την καταπολέμηση της φτώχειας, δεν πρόκειται να πετύχουμε το στόχο που έχουμε θέσει να μειώσουμε δηλαδή τους ανθρώπους εκείνους που εκτίθεται στον κίνδυνο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού κατά 20 εκατομμύρια μέχρι το 2020. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να αντιμετωπίσουμε τις πτυχές που έχουν να κάνουν με το φύλλο όσον αφορά το ζήτημα της φτώχειας. Πρέπει να δεσμευτούμε λοιπόν για τους στόχους αυτούς της στρατηγικής 2020 και να έχουμε μια σφαιρική στρατηγική μείωση της φτώχειας επικεντρώνοντας το ζήτημα του φύλου. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να πούμε ότι υπάρχει πλέον ένας έντονος γυναικείος χαρακτήρας όσον αφορά το φαινόμενο της φτώχειας. Έχω έρθει σε επαφή με πάρα πολλές ομάδες της κοινωνίας, έχω συνεργαστεί με τους συναδέλφους από την Επιτροπή Απασχόλησης. Η έκθεση της Επιτροπής αυτής αναφέρεται κυρίως στο ζήτημα της ενεργειακής ένδυας. Μολονότι το ζήτημα αυτό είναι πολύ σημαντικό και πλήττει ιδιαίτερα και τις γυναίκες, θεωρώ ότι η δική μας η θα πρέπει να αναφερθεί σε επιπλέον διασυνδεδεμένα στοιχεία που έχουν να κάνουν με τη φτώχεια, όπως για παράδειγμα το ζήτημα των αποδοχών. Νομίζω ότι θα πρέπει να αναφερθούμε στον διατομιακό χαρακτήρα, χαρακτήρα των πτυχών της φτώχειας, που σχετίζονται με το φύλλο, να μην ασχολούμαστε μόνο με την ηλική φτώχεια και ένδια, αλλά να δούμε πραγματικά τι χρειάζονται ιδίω οι γυναίκε για να μπορούν να συμμετέχουν πιο ενεργά στην κοινωνία και να μπορούν να ενσωματώνονται εκ νέου οικονομικά και κοινωνικά στην κοινωνία. Έχω έρθει σε επαφή με διάφορου οργανισμού, όπω σα είπα, οι οποίοι μου έχουν πει ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό γυναίκε να μπορούν να ζουν με αξιοπρέπεια. Ξέρετε ότι οι γυναίκε κινδυνεύουν ιδιαίτερα από τη φτώχεια και από τον κοινωνικό αποκλεισμό, δυσανάλογα επίση έχουν πληγεί από την κρίση και τι πολιτικέ λιτότητο. 23,6% των ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση πλήττονται από τη φτώχεια, ενώ 25,4% των γυναικών κινδυνεύουν να πληγούν από τη φτώχεια. 22% οι άνδρες, 24% οι γυναίκες το 2010. Ήταν τα αντίστοιχα ποσοστά. Βλέπετε λοιπόν ότι είχαμε και αύξηση τα τελευταία πέντε χρόνια. Επίσης, ε, οι γυναίκες είναι πιο ευάλωτες από τις περικοπές στις δημόσιες υπηρεσίες και μπορεί πολύ πιο εύκολα να βρεθούν σε επισφαλείς θέσεις απασχόλησης. Όσον αφορά την ενεργειακή ένδια, ένα 17% των μονεγωικών οικογενειών με αρχηγό ουσιαστικά γυναίκες δεν καταφέρνουν να έχουν πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες όπως η θέρμανση. Βλέπαμε και κάποια περαιτέρω αριθμητικά δεδομένα και βλέπαμε ότι ε, χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου έχουμε πολλούς κρύους ε, χειμώνες, είναι χώρες όπου οι γυναίκες εκτίθενται περισσότερο σε σχέση με τις μεσογειακές χώρες. Στις μεσογειακές όμως χώρες έχουμε και εκεί τεράστια προβλήματα με την ε, θέρμανση για παράδειγμα. Επομένως δεν μπορούμε να πούμε ούτε και για τα ζητήματα αυτά ότι οι χώρες, ε, οι βόρειες πλήττονται περισσότερο όσον αφορά για παράδειγμα την ενεργειακή ένδυα. Το ζήτημα αυτό της ε, θέρμανσης των σπιτιών πραγματικά αντικατοπτρίζει τα γενικότερα προβλήματα που όλες οι γυναίκες παντού στην Ευρώπη αντιμετωπίζουν. Επίσης έχουμε διακριτική μεταχείριση όσον αφορά τις γυναίκες, γυναίκες που βρίσκονται σε συγκεκριμένες κατηγορίες όπως πρόσφυγες, άτομα με ειδικές ανάγκες, κοινότητες των δρομά, Έχουμε συγκεκριμένες ομάδες που είναι ακόμα πιο ευάλωτες και για τις οποίες χρειαζόμαστε συγκεκριμένες πολιτικές και οι πολιτικές αυτές θα πρέπει να ενταχθούν στις εθνικές στρατηγικές μείωσης της φτώχειας. Τώρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να έχουμε μεγαλύτερη πολιτική συνεκτικότητα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη. Θεωρώ ότι είναι παράλογο να προωθούμε ένα γενικότερο κλίμα δημοσίων περικοπών και λιτότητας που αυξάνει από τη μία πλευρά τη φτώχεια και από την άλλη να λέμε ότι θέλουμε να έχουμε περισσότερες κοινωνικές πολιτικές. Νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο θα πρέπει να έχει μια, ένα πιο έντονο κοινωνικό χαρακτήρα και κοινωνικό επίσης χαρακτήρα θα πρέπει να έχουν και ειδικέ αναχώρα συστάσεις του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας έχει προτείνει μια κοινωνική Ευρώπη τριπλού Α. Πρέπει πραγματικά να δούμε όμως σε τι αντιστοιχεί αυτό και αν πραγματικά οι προθέσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι φιλόδοξες. Ερχόμενοι σε επαφή με οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών, συντοποίησε ότι υπάρχουν συγκεκριμένα ζητήματα τα οποία πρέπει να φυγούν. Πραγματικά είδα τα πράγματα με μία φρέσκια ματιά, δεν είχα προσεγγίσει το ζήτημα αυτό στο παρελθόν, χρειάστηκε λοιπόν να μελετήσω λίγο το ζήτημα αυτό. Υπάρχει ένα πρόβλημα με, τον, με τη χρησιμοποίηση του όρου νοικοκυριό γιατί αντιμετωπίζεται από όλους τους δείκτες όρος αυτός με τρόπο εντελώς ομοιόμορφο, ενώ το ένα νοικοκυριό διαφέρει πάρα πολύ από το άλλο. Πολύ συχνά στα πλαίσια των λεγόμενων νοικοκυριών έχουμε πολύ άνηση κατανομή των εισοδημάτων. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να υπάρχει μία εξατομίκευση των δεδομένων που χρησιμοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε να φαίνεται περισσότερο η περίπτωση εκείνη των γυναικών που ζουν μόνες τους ή είναι υπεύθυνε για μία οικογένεια. Είναι πολύ σημαντικό επίσης στα πλαίσια των κρατών μελών να μπορούμε να επικεντρωθούμε περισσότερο στο πόσο ευάλωτες είναι οι γυναίκες καταναλωτέ. Επίσης οι εθνικές πολιτικές όσον αφορά την ενεργειακή, τις ενεργειακές επιδόσεις θα πρέπει να επικεντρωθούν σε κάποιους ευάλωτους καταναλωτές όπως οι γυναίκες, οι οποίες είναι θύματα πολλαπλών διακρίσεων. Χρειαζόμαστε περισσότερα δεδομένα όσον αφορά τις άστεγες γυναίκες και τη διασύνδεση που υπάρχει ανάμεσα στην τιμή των ακινήτων, τα εισοδήματα, καθώς επίσης και την κατάσταση την επαγγελματική στην οποία βρίσκονται οι γυναίκε. Πολλέ φορέ οι άστιγε γυναίκε δεν περιλαμβάνονται καθόλου στα επίσημα αριθμητικά δεδομένα. Δεν καταφέρνουμε να τι εντοπίσουμε, δεν τι βλέπουμε καν στου δρόμου. Πολύ συχνά δεν προσπαθούν καν να υποφεληθούν από τις διάφορε δημόσιε υπηρεσίε που υπάρχουν για του ε, άστεγους δεν εμφανίζονται λοιπόν καθόλου στα επίσημα δεδομένα. Θα πρέπει επίσης να καταλήξουμε σε κάποιες ευρωπαϊκές ε, συστάσεις όσον αφορά τους ε, αξιοπρεπείς ε, μισθούς, όσον αφορά το επίπεδο χρέους των γυναικών, όσον αφορά την φορολογία που πλήττει ή επηρεάζει τις γυναίκες. Πρέπει να κλείσουμε επίσης το μισθολογικό χάσμα και την ανισότητα που υπάρχει μεταξύ ανδρών και γυναικών. Επίσης, πολλές ε, οργανώσεις γυναικών θα πρέπει όλο και περισσότερο σε όλα τα επίπεδα να μπορούν άμεσα να συμμετέχουν. Γίνονται επίσης κάποιες πολύ άλλες πιο συγκεκριμένες συστάσεις, τις οποίες θα ήθελα να κάνω στα πλαίσια της έκθεσης αυτής. Δεν έχω τον απαραίτητο χρόνο. Το βασικό μήνυμα πάντως είναι ότι η φτώχεια έχει έναν έντονο διατομιακό χαρακτήρα που συνδέεται με το φύλλο και πολλές φορές περνάει από τη μία γενιά στην άλλη η φτώχεια αυτή αν δεν αντιμετωπιστεί πολύ νωρίς. Καταλαβαίνετε ότι όταν πλήττονται για παράδειγμα οι γυναίκες από τη φτώχεια, πολύ σύντομα και τα ίδια τα παιδιά τους θα πλήττονται από τα ίδια επίπεδα φτώχειας. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει για όλα αυτά τα ζητήματα να προτείνουμε λύσει και περιμένω και τις δικές σας τις προτάσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστούμε κύριε Ward. Υπάρχει κάποιος, ε, κάποια συνάδελφος ε, που θα ήθελε το λόγο. Είστε όλες 100% ικανοποιημένες. Α, εσείς. Α, συμφωνώ με αυτά που είπε η Τζούλη μόλις τώρα, πόσο δύσκολο είναι να έχουμε αριθμητικά στοιχεία, στατιστικές ε, για τις γυναίκες αυτές. Ε, γίνονται εξαρτώμενα άτομα λόγω της στόχης οι γυναίκες και οι άστεγες ε, τι σημαίνει να είναι κανείς άστεγος, δεν έχει σπίτι, δεν έχει στέγη. Πέραν αυτού δεν έχει ένα ασφαλή, ασφαλή χορό που μπορεί να αφήσει τα πράγματά του, ε, να νιώσει ασφαλής. Ε, και γίνονται εξαρτώμενα τα άτομα, ε, οι γυναίκες αναγκάζονται να εκδοθούν Ε, ασχολήθηκα στην ε, Οξφορδή με αυτές τις ε, γυναίκες ε, και μου είπανε ότι μπορείς να, τις, να ξέρεις τι, ότι κάποιος είναι αστεγός διότι δεν κοιμάται, κάθεται ξύπνιος γιατί είναι ασφαλέστερο. Και μόνο όταν κοιμούνται μπορεί κάποιος να τις καταμετρήσει. Ε, και υπάρχει λοιπόν αυτό το διπλό μειονέκτημα πέρα από τη φτώχεια όταν δεν έχουν ε, σπίτι ε, είναι πολύ αρνητικότερο ο αντίκτυπο και θα πρέπει να καταλήξουμε ίσω σε έναν ορισμό και να ενσωματώσουμε κάτι μέσα στην έκθεση. Κυρία Βυσνιεύσκα, ευχαριστώ. Είναι πολύ δύσκολο το όνομά μου, το παραφύρετε συστηματικά. Ελπίζω κάποια στιγμή να το προφέρετε στο μέλλον σωστά. Είναι πάρα πολύ ε, ενδιαφέρον αυτό το πρόβλημα που πραγματεύεστε μέσα στην έκθεση, πώς μπορούμε να καταπολεμήσουμε τη φτώχεια ενώ ταυτόχρονα αυξάνονται οι δαπάνες στα νοικοκυριά. Δύσκολα κανείς μπορεί να αγνοήσει το ότι ε, αυξάνεται και ο αριθμός των ενεργειακά αποξενωμένων, αποκλεισμένων. Είναι αυξανόμενο, ε, ε, είναι αυξανόμενος ο αριθμός των ανθρώπων που δεν μπορούν πλέον να πληρώσουν το ηλεκτρικό ρεύμα. Δεν έχουν θέρμανση γιατί δεν έχουν χρήματα για να πληρώσουν. Θα πρέπει αυτό να συμπεριληφθεί στην πολιτική καταπολέμηση τη φτώχεια. Επίσης να επικεντρωθούμε ε, στο θέμα τη φτώχεια των μονογονεϊκών οικογενειών ή ε, το αντίστροφο των ε, πολυμελών οικογενειών. Από πού προκύπτει το φαινόμενο της στόχιας, από την φορολογική πολιτική, στην οικονομική πολιτική χρειαζόμαστε ρυθμίσεις τομεακού χαρακτήρα να εξασφαλίσουμε πρώτα απ' όλα καθολική πρόσβαση στο ηλεκτρικό ρεύμα. Και αυτό δεν σχετίζεται υποχρεωτικά με τη διάσταση του φύλου. Αναφερθήκατε στους αστέγους και καλά κάνατε. Γίνονται διαφανείς, αόρατοι αυτοί οι άνθρωποι κάποια στιγμή. Δηλαδή δεν τους προσέχουν οι συνάνθρωποι τους. Ίσως θα έπρεπε να εξετάσουμε και κάποιες διαστοτικού τύπου λύσεις. Οι φτώχες της πολυμελής οικογένειας δείχνει ότι αποτυγχάνουμε ως τις πολιτικές που εφαρμόζουμε και από ό,τι φαίνεται το βασικότερο πρόβλημα είναι ακριβώς η φτώχεια στις πολυμελείς οικογένειες και πλήττει πολλά κράτη-μέλη. Η οικογενειακή πολιτική, η κοινωνική μας πολιτική πόρο απέχουν από την τελειότητα και αποτυγχάνουν στο να αντιμετωπίσουν αυτό το φαινόμενο. υποστήριξη προς τις μονογονεϊκές οικογένειες, άλλο σημαντικό ζήτημα. Επίσης, θα πρέπει να έχουμε κατά νου πως τα προγράμματα δεν θα πρέπει να ε, ευνοούν ε, τα εικονικά διαζύγια για να έχουν ευνοϊκότερες επιδοτήσεις, ε, διότι και αυτό συμβαίνει σε πάρα πολλές χώρες, για να παίρνουν περισσότερα και καλύτερα επιδόματα, τείνουν να επιλέγουν το διαζύγιο οι γονείς για να μπορέσουν να εποφεληθούν από τις ευνοϊκότερες κοινωνικές ρυθμίσεις. Ευχαριστώ πολύ κυρία Φυσνέσκα. Ευχαριστώ πολύ, το είπατε. Κύριε Σεπάστια, θα ήθελα να πω δύο λόγια για το θέμα του καλού καιρού στις χώρες τη Μεσογείου. Βέβαια εξαρτάται αυτό, ξέρετε. Άλλο στην παραλία, η πρόεδρος μένει στην Ισπανία, που υποτίθεται είναι ζεστή χώρα, αλλάζει στο κέντρο της χώρας όπου οι χειμώνες είναι βαρύς. Σε διαβεβαιώνω. Στην Πορτογαλία, την Ισπανία, την Ιταλία, μην ξεχνάτε ότι έχουμε και πολλά κτίρια που χτίστηκαν είτε τους προηγούμενους αιώνες είτε στη δεκαετία του 70 και του 80 που δεν ε, συνάδουν με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και έτσι πώς θα ζεστάνεις το σπίτι η ενεργειακή δαπάνη είναι μεγαλύτερη ίσω κάποια στιγμή και από αυτήν του βορρά. Δηλαδή μπορεί να κάνει 10 βαθμούς έξω και να κάνει και 10 και μέσα στο σπίτι. Το οποίο σημαίνει ότι κάνει κρύο για μια μέση οικογένεια. Το λέω αυτό γιατί μερικοί νομίζουν ότι στο Νότο εμεί δεν έχουμε τέτοια προβλήματα. Ε, ενδιαφέρον πάντως αυτό που είπατε. Ευχαριστώ, συγχαρητήρια. Muchas eh, Πολύ ωραία. Η κυρία Word νομίζω θέλει να κλείσει, αν δεν, υπάρχει κάποιος άλλος. Ναι. Κυρία Word. Ευχαριστώ για τα σχόλια. Βλέπω υπάρχει ευρεία υποστήριξη, εξαιρετικά. Αυτό κάνει πιο εύκολη τη δουλειά μου. Κάθριν, ευχαριστώ, διότι τόνισες για άλλη μια φορά το θέμα των αστέγων. θα ήταν ίσως χρήσιμο να ξέρετε με ποιους μίλησα, με ποιες οργανώσεις, όπου πήρα τα στοιχεία. Μιλήσαμε για το Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Φτώχειας, την Ευρωπαϊκή Διακονία, με την οποία είχαμε μια εξαιρετική συνάντηση χθε. Είναι μια θρησκευτική οργάνωση, η οποία υποστηρίζει ε, ανθρώπους σε ακραία ένδια. Γνωρίζουν το θέμα, γνωρίζουν τους ανθρώπους, ένα προς έναν κάνουν σπουδαία δουλειά σε διάφορες χώρες και μας έδωσαν πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Μιλήσαμε με, με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Ισότητας των Φύλων και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την απόδοση. Εκεί μίλησα για συγκεκριμένα θέματα σχετικά με τα κτίρια, τα, τα σπίτια, το πώ έχουν χτιστεί. Ξέρω ότι μάλιστα την κατάσταση στην Πορτογαλία, γιατί πέρασα τον Δεκέμβριο δύο εβδομάδε στα πορτογαλικά βουνά σε ένα σπίτι που ήταν ακριβώς αυτό όπως το περιγράψετε. Και εγώ περίμενα ότι θα πάω στο Νότο να ζηταθώ και είναι το αντίθετο. Λοιπόν, το τονίζω αυτό, διότι εμεί στο Βορρά πιστεύουμε ότι μόνο εμεί κρυώνουμε. Είναι και για εσά το πρόβλημα. Ε, οι στατιστικέ πολλέ φορέ δεν το αποτυπώνουν. Και μιλούμε επίση για το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αστέγων. Ε, θέλω να πω ότι μίλησα με πάρα πολλέ οργανώσει τη κοινωνία των πολιτών, να το ξέρετε αυτό και με πολλές οργανώσεις αρρωγής που μου παρέσχουν τα σχετικά στοιχεία όσον αφορά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού, την μεταβολή του κλίματος κλπ. Για μένα δεν είναι είτε το ένα είτε το άλλο. Θα λέω ότι είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο με την εξής έννοια. Ήμουν σκιώδης σε έκθεση Μόνικα Βάνα έκθεση αυτή τη Επιτροπή σχετικά με τι πράσινε θέσει εργασία για τι γυναίκε. Λοιπόν, στην Επιτροπή μα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα ολιστικά. Γιατί έχουμε πολλά ζητήματα, όπω η φτώχεια, μεταξύ άλλων βεβαίω. Και έχουμε και προβλήματα σχετικά με την αξιοπρέπεια των γενικών, των γυναικών. Ε, έχουμε το θέμα τη μεταβολή του κλίματο και ένα σωρό άλλα πράγματα. Λοιπόν, δεν έχει πολύ νόημα να μιλήσουμε για τα ορεικτά καύσιμα και να αποκλείσουμε τη μία την άλλη ενεργειακή πολιτική επειδή οι γυναίκες δεν μπορούν να πληρώσουν το ρεύμα. Όλα αυτά χρειάζονται μια την αλλη ενεργειακη πολιτικη επειδη οι γυναικε δεν μπορουν να αντιμετώπιση για να επικεντρωθούμε στη ρίζα, στην αιτία του προβλήματος. Και ούτω ή άλλω αυτά αφορούν και τις επόμενε γενναίε. Γι' αυτό λέω και τονίζω για μια φορά την ανάγκη ολιστικής προσέγγιση. Το θέμα τη απόδοση λοιπόν είναι πολύ σημαντικό. Αυτό είναι τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε. Ύστερα η λιτότητα είχε ως κύριο θύμα τις γυναίκες. Οι γυναίκες δηλαδή εν τέλει έχουν τις περισσότερες δυσκολίες να, από το να πληρώσουν το ρεύμα μέχρι οτιδήποτε άλλο λόγω της λιτότητας. Εγώ στην, νοτιο, στην βορειοδυτική Αγγλία και ξέρω ότι στην εκλογική μου περιφέρεια υπάρχουν πολύ φτωχοί. Βέβαια, φτωχοί και προηγουμένω, αλλά οξύθηκε περισσότερο το φαινόμενο μετά. Μετά δηλαδή την επέλευση τη κρίση. Αυτά νομίζω απήντησα στα περισσότερα τουλάχιστον. Σε αυτά θα περιοριστώ. Ευχαριστώ πολύ για την υποστήριξη. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, η προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών είναι η 10η Δεκεμβρίου, 12 το μεσημέρι. Μετά στις 28 Ιανουαρίου θα ψηφίσουμε στη δική μας την Επιτροπή και στη συνέχεια στις 17 Φεβρουαρίου θα διεξαχθεί ψηφοφορία στην Επιτροπή Απασχόλησης, η οποία είναι η καθήλυνα αρμόδια. Ολοκληρώνουμε λοιπόν και αυτό το σημείο στη μερίσια διάταξη. Περνάμε τώρα στις ψηφοφορίες. Ας διακόψουμε για ένα-δύο λεπτά, προκειμένου να καθίσετε όλοι, να βρείτε τις κάρτες ψηφοφορίας. Okay. Eh, λοιπόν, νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε τώρα. Ξεκινάμε λοιπόν με την ε, γνωμοδότηση της κυρίας Μπιόρκα, εφαρμογή των συστάσεων του Κοινοβουλίου του 2010 σχετικά με τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την εταιρική ευθύνη. Ξεκινάμε λοιπόν, αν είστε όλοι έτοιμοι. Τροπολογία 16 πέρα. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονική παρήθευση. Παρακαλώ, άρχιτη ψηφοφορία. Τροπολογία 16. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 17 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 32, συγγνώμη, 19 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 21 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 20 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 22 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 23 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 6 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 33 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 34 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 35 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές ηλεκτρονική επαλήθευση λοιπόν για την τροπολογία 35 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Και εγκρίνεται. Τροπολογία 36 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 37 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 39 υπέρ. Έχουμε προφορική τροπολογία για την 39, με ενημερώνουν. Κυρία Μπίαρντερ, έχετε κάποια προφορική τροπολογία, θέλετε να διαβάσετε. Πρόκειται για μια διόρθωση που έγινε στη μετάφραση. Λέγεται παρατηρεί ότι η διάσταση του φύλου στην εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι πλήρως ενσωματωμένη στη στρατηγική για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών. Να λέγεται ανταυτού ότι η στρατηγική τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών δεν έχει λάβει δεόντως υπόψη τη διάσταση του φύλου στην εμπορική πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολύ ωραία λοιπόν συμπεριλαμβάνουμε αυτή την προφορική τροπολογία υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 40 υπέρ, κατά, αποχές, ηλεκτρονική επαλήθευση για την τροπολογία 40, άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 42 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 4 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ψηφίζουμε τώρα ηλεκτρονικά τελική ψηφοφορία το κείμενο όπως τροποποιήθηκε άρτη ψηφοφορία Πέρας. Και εγκρίνεται. 15 υπέρ, 8 κατά και 2 αποχές. Συγχαρητήρια λοιπόν στην κυρία Μπιόρκ. Y τώρα την ε, ψηφοφορία για τη γνωμοδότηση όσον αφορά την εφαρμογή και επανεξέταση στρατηγικής Ευρωπαϊκής Ένωσης Κεντρικής Ασίας 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 21 έχει αποσυρθεί 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 4 υπέρ συμβαστική κατά αποχές εγκρίνεται 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές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 εγκρίνεται. 6 υπέρ σε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα της 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα της 6 υπέρ κατά αποχές. Κουραστήκαμε λίγο νομίζω. Δεν σηκώνετε αρκετά τα χέρια σας νομίζω. Δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 6 υπέρ παρακαλώ. Πολύ καλύτερα τώρα. Κατά.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 Πολύ ωραία. Ηλεκτρονική λοιπόν ψηφοφορία για το κείμενο που τροποποιήθηκε. Άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Καταπληκτικά 25 υπέρ, 2 κατά και μία μόνο αποχή. Συγχαρητήρια λοιπόν στην κυρία Γκέρλινγκ. Bueno, pues ya hemos dado un Ωραία. Τώρα ε, κάναμε και ένα μικρό διέλματάκι. Μπορούμε να προχωρήσουμε τώρα. Θα αρχίσουμε με το σημείο 7. Έκθεση για τις γυναίκες απασχολούμενε ω οικιακές βοηθοί και ω προσωπικό φροντίδες εξαρτώμενων ατόμων. Η συγγήτριά μας είναι η Κωνσταντίνα Κούνεβα. Ε, γνωμοδότηση προς Επιτροπή Απασχόλησης. Έχετε το λόγο, κυρία Κούνεβα, για την παρουσίασή σας και μετά θα γίνει συζήτηση. Ευχαριστώ πάντα. Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, αρχικά να σας ευχαριστήσω όλους για τις τροπολογίες που καταθέσατε. Διαπίστωσα πως σε πολλές από αυτές οι σκέψεις μας ήταν κοινή, κάτι που με χαροποίησε ιδιαίτερα. Θα ήθελα όμως να καταλάβω γιατί κάποιοι συνάδελφοι δεν θέλουν νομοθετικέ πρωτοβουλίε που να ρυθμίζουν αυτές τι κατηγορίες εργαζομένων, δεδομένου ότι μιλάμε για ανθρώπους που έχουν την χαμηλότερη προστασία, πώ έχουμε στο μυαλό μας να του προστατεύσουμε. Αρκεί να σας πω πως η απόφαση για την δημιουργία πλατφόρμα για την καταπόλεμηση της αντιότητας που ψηφίστηκε πριν από λίγο στην Επιτροπή Απασχόληση, περιλαμβάνει αυτό το τύπο του εργαζομένου. Κάποιοι συνάδελφοι είναι αντίθετοι ακόμα και με την καλύτερη εφαρμογή των κανόνων προστασίας που ήδη υπάρχουν. Πώς είναι δυνατόν και γιατί το ζητάμε αυτό. Σας αφήνω να σκεφτείτε τα παραπάνω ερωτήματα και να προχωρήσω και να σταθώ σε μερικέ από τι τροπολογίε τι οποίε θα ήθελα να συζητήσουμε. Το πρώτο σημείο στο οποίο θα ήθελα να αναφερθώ είναι η τροπολογία 78 της κυρίας Μπλίνκεβιτσιώτε, όπου αναφέρει πω θα πρέπει να υπάρχει αναγνώριση τη αξία τη οικιακή εργασία και φροντίδα. Σε αυτή τη σκέψη συμφωνώ εν μέρη. Δεν αρκεί να αναγνωρίζουμε την αξία των παρεχόμενων υπηρεσιών. Χρειάζεται να αναγνωρίσουμε και να προχωρήσουμε με νομοθεσία που αφορά στην ρύθμιση του επαγγέλματο αυτού. Σε ό,τι αφορά τι τροπολογίε 93 και 94, με τι οποίε ζητείται η διαγραφή τη προστασία να συντάξει μια έκθεση νομοθετική πρωτοβουλία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δυστυχώ διαφωνώ. Αν δεν κάνουμε εμεί το πρώτο βήμα. Αν δεν δώσουμε την απαραίτητη όθηση για να ξεκινήσει η διαδικασία ρύθμισης του φαινόμενου της οικιακής εργασίας και φροντίδας, τότε ποιος ακριβώς είναι ο ρόλος μας. Να επαναλαμβάνουμε ευχολόγια. Γι' αυτό σας καλώ να σκεφτείτε ξανά για ποιο λόγο συντάσσουμε την έκθεση αυτή. Η τροπολογία 107 θεωρώ πως αναφέρει σε ένα σημαντικό βήμα για να προχωρήσουμε στην προστασία των οικιακών εργαζομένων και των προσωπικών φροντίδας είναι ο κανονικός διάλογος. Και η τροπολογία αυτή είναι σε πολύ καλή κατεύθυνση. Σε ό,τι αφορά τη διάσταση των μεταναστών οικιακών εργαζομένων, τροπολογία 136, διατυπώνει μια πολύ καλή πρόταση που συμπληρώνει αυτή την κα... που κρατέσαμε και εμείς αρχικά. Επίσης, χάρηκα ιδιαίτερα με τις τροπολογίες 140, 141 και 142 και 143, όπου προτείνεται να συντάξει η Κομισιόν μια έκθεση που θα αποτυπώνει πόσο μεγάλη είναι η συνεισφορά και η αξία της προσφερόμενη οικιακή εργασία και φροντίδα. Και θεωρώ πω, όταν η έκθεση αυτή ολοκληρωθεί θα φαίνεται εκτός από την ε, κοινωνική αξία της εργασίας αυτής πόσο συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη κάτι κοινωνίας. Η τροπολογία 148 είναι καλή και γενικά συμφωνώ μαζί της. Ωστόσο, Νομίζω ότι θα πρέπει να πάμε ένα βήμα πίσω. Πριν ζητήσουμε από τους εργαζόμενους που θέλαμε να απασχολήσουμε σπίτια μας να έχουν συγκεκριμένα προσόντα, θα πρέπει εμείς να φροντίσουμε να έχουμε ένα σύστημα που θα αναγνωρίσει το επάγγελμα, θα πιστοποιεί τις δεξιότητες που έχουν εργαζόμενοι, αλλά και θα τους επιτρέπει να εκπαιδεύονται και να εξελίσσουν τα προσόντα τους αυτά. Ακόμα πολύ ενδιαφέρουσα είναι η τροπολογία 159 για την προστασία του οικιακού προσωπικού στις διπλωματικές οικίες για τις οποίες δεν σας κρύβω είχα συναντήσει αρκετές φορές περιπτώσεις κατά την προετοιμασία της έκθεσης όπου αναφερόταν περιπτώσεις κακοποίησης και εκμετάλλευσης διάφορων μορφών. Σε ό,τι αφορά τις τροπολογίες του κυρίου Ουρτασούν. Τον ευχαριστώ πολύ που έδωσε τόσο βάρος στο κομμάτι του τράφικινγκ ένα φαινόμενο με ξεκάθαρη φιλητική διάσταση και ακόμα συνδέεται με πολλές μορφές αναγκαστικής εργασίας και βίας σεξουαλικής, λεκτικής και άλλων μορφών. Σε ό,τι αφορά τις τροπολογίες 162 που αφορούν την ομοθεσία που πρέπει να εφαρμόσουν τα κράτη-μέλη δεν αρκεί να κάνουμε άλλη μια σύσταση ούτε να ζητήσουμε πρωτοβουλίες. Είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να πιέσουμε. Η σκέψη της κυρίας Φάρεγκουτ και Ματέρα είναι καλή, αλλά νομίζω πως είναι λίγο επιδερμητική. Κλείνοντας, να συναψίσω λέγοντας πως πολλές τροπολογίες θα πρέπει να συμπεριφθούν σε συμβατικές κατός αφορούν ζητήματα που θίγονται ήδη στην έκθεση, αλλά προσθέτουν και άλλα στοιχεία πολύ χρήσιμη για την ακόμα καλύτερη προστασία των εργαζομένων σε αυτούς τους τομείς. Τέλος, θα τα ζητήσω για άλλη μια φορά να στηρίξουμε την έκθεση αυτή και να δουλέψουμε μαζί για να κάνουμε ξεκάθαρο πως όσοι ζουν στα σπίτια μας φροντίζουν τους γονείς και τα παιδιά μας, καταρίζουν, μας δίνουν το χρόνο να δουλέψουμε και να απολαμβάνουμε την κοινωνική μας ζωή. Αυτή η πολύτιμη κατηγορία εργαζομένων δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται σαν εργατικό δυναμικό β' κατηγορίας και δεν πρέπει να πέφτουν θύματα διάκρισης λόγω του φίλου τους. Και αυτά πρέπει να γίνει μια και καλή ξεκάθαρο. Εμονή και αποφασιστικότητα. Με κάτι μας πράξει με κάτι μας λέξη. Εδώ μέσα πρέπει να δείχνουμε τις, τις γυναίκες και προκειμένου τις οικιακά εργαζόμενες ότι δεν τις έχουμε εγκαταλείψει. Σε ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε, κυρία Κούνεβα. Θα αρχίσουμε τώρα τη συζήτηση. Ποιος θα ήθελε το λόγο, παρακαλώ. Μίλνα, Αγιωτό. Ας αρχίσουμε τότε. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Κούνεβα για τη δουλειά που έχει κάνει και να σα ενημερώσω ότι θέλουμε να ενισχύσουμε τρεις πτυχές που ήδη αναφέρεται στην έκθεση μέσα από τις τροπολογίες μας, τη, διάσταση της εκμετάλλευσης. Ε, ο τομέας των οικιακών βοηθών όπου η πλειοψηφία ε, είναι γυναίκες, ε, δυστυχώς δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για την εκμετάλλευση. Είναι μια γκρίζα ζώνη δυστυχώς και η εκμετάλλευση ορισμένες φορές δεν εκλαμβάνεται ως παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και γι' αυτό χρειαζόμαστε αποτελεσματικότερη ισχυρότητα περισσότερη προστασία των οικιακών βοηθών ε, και για την αδήλωτη εργασία και για του πολίτε Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, δεύτερον, η σχέση με τη μετανάστευση, ε, διότι είναι πολλέ οι μετανάστε που εργάζονται σε αυτό το τομέα και εκτίθενται σε ιδιαίτερο κίνδυνο εκμετάλλευση. Επίση, η αδήλωτη εργασία του έχει ω αποτέλεσμα ότι δεν υπερασπίζονται τον εαυτό του και δεν φοβούνται ότι θα απελαθούν, θα εντοπιστούν θα απελαθούν και γι' αυτό δεν εκδηλώνονται. Τρίτον, η αναγνώριση αυτού του επαγγελματικού τομέα ή γενικότερα η επαγγελματικοποίησή του. Δηλαδή, θεωρούμε ότι ο τομέα αυτό μπορεί να δημιουργήσει θέσει εργασία, ανάπτυξη και μπορεί να είναι μέρο ενό κοινωνικού και οικονομικού μοντέλου. Μπορούμε έτσι να καταστήσουμε αυτόν τον τομέα ελκυστικότερο, να αναβαθμιστεί η ποιότητα των υπηρεσιών και όλα αυτά μέσα από την αναγνώριση των επαγγελματικών υπηρεσιών που παρέχονται. Σίγουρα θα είναι ε, καρποφόρα η συνεργασία μας και θα μπορέσουμε να έχουμε στο τέλος μια πολύ καλή έκθεση. Σας ευχαριστούμε ε, κυρία Μίλνερ και κυρία Κοράτσια Μπίλτ. Ευχαριστώ. Εγώ τοποθετούμε από πλευρά τη Ρόζα Εστορία, ε, που είναι η συγγήτρια, η συγγήτρια του ΕΛΚ, η οποία όμω δυστυχώ δεν μπορούσε να παρευρεθεί σήμερα. Ευχαριστεί την συγγήτρια, διότι θέτει αυτό το τόσο σημαντικό ζήτημα προς εξέταση ε, πολλές φορές ε, δεν ε, παραγνωρίζεται η σημασία της πολιτική συζήτηση να αναγνωριστεί λοιπόν η αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα των οικιακών βοηθών και του προσωπικού φροντίδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση πως επιτοπλίστων είναι μετανάστριες γυναίκες είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να εκδηλώσουμε ε, πλήρη υποστήριξη ε, για την καταπολέμηση της εκμετάλλευσης, ε, της παράνομης απασχόλησης και για να υποστηρίξουμε τη μετάβαση από την αδήλωτη στην δηλωμένη εργασία. Ίσως χρειαστεί μια μελέτη για να γίνει σύγκριση ανάμεσα στις βέλτιστες πρακτικές των κρατών μελών. Θεωρεί επίσης η κυρία Ρόζα Ιστορίας. Αρχίζω με τα θετικά σημεία, Πρόεδρε. Ε, για το θέμα ε, του σημείου 11 για την υποχρέωση ενημέρωσης, το 19 για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού. Εκεί θα ενθαρρύνουμε και θα καλέσουμε τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν τις ε, απαιτούμενες πολιτικές ε, κατά της ε, κοινωνικής αποξένωσης. Επίσης, το σημείο για την εγκατάλειψη της εκπαίδευσης για να επανενταχθούν τα παιδιά στο εκπαιδευτικό σύστημα. Τώρα, ποιο είναι το προβληματικό σημείο, πολύ προβληματικό μάλλον για το ΕΛΚ, είναι το ζήτημα ότι για το εργατικό δίκαιο δεν έχουμε καμία αρμοδιότητα. Δηλαδή, η έκθεση αυτή πραγματεύεται σημεία που εκφεύγουν τι αρμοδιότητε μα. Είναι πολύ καλό λοιπόν να το θέτουμε προς και προ εξέταση το ζήτημα. Αυτό είναι ένα πράγμα, αλλά πολύ διαφορετικό είναι να ζητούμε ε, νομοθετική ρύθμιση από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω στην παράγραφο 2 και 3. Δηλαδή, τονίζουμε την ανάγκη να υπάρξει ρύθμιση για ε, τι οικιακέ βοηθήσει και το προσωπικό φροντίδα και καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ασκήσει το δικαίωμα πρωτοβουλία και να καταθέσει νομοθετική πρόταση. Και το ίδιο και στην επόμενη παράγραφο. Ζητούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να νομοθετήσει και θεωρούμε ότι δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητά μα κάτι τέτοιο. Η σχεδόν συγκίτρια του ΕΛΚ είναι επίσης κατά ε, της ε, ε, συγκρότησης ενός παρατηρητηρίου σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για το ζήτημα αυτό ε, στο σημείο 15 πάλι για λόγους επικουρικότητας παράγραφοι 12 και 13 για το ρόλο των συνδικαλιστικών οργανώσεων και αυτό είναι εθνικό ζήτημα Επίσης, η κοινοποίηση της σύμβασης του Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που είναι αυτό, είναι στο σημείο 6 και το τελευταίο σημείο είναι το 22. Ζητά από τα κράτη μέλη να ελέγξουν το θέμα των φορολογικών ελαφρύνσεων και των επιδομάτων και αυτό είναι θέμα επικουρικότητας. Αυτά λέει η συνάδελφος Ρόζα και εγώ από πλευράς μου να προσθέσω ένα σύντομο σχόλιο. Εγώ θεωρώ ότι ε, ε, είναι μια μικρή ανακολουθία, διότι δηλαδή η αριστερά προσπαθεί πάντοτε να καλέσει την Ευρωπαϊκή Ένωση να ε, παραβιάσει το, το αποκλειστικό δικαίωμα των ε, κρατών μελών και την αρμοδιότητά τους. Δεν είναι ότι δεν είμαι ε, υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν είναι αυτό το ζήτημα, όμως υπάρχουν το τομεί όπω η ασφάλεια που χρειάζεται συνεργασία διότι είναι διατομεακά τα ζητήματα και υπάρχουν άλλα ζητήματα που είναι ξεκάθαρα εθνική αρμοδιότητα ε, και θεωρώ ότι είναι ασυνεπέ από πλευρά αριστερά να ζητά ε, ενωσιακή ρύθμιση σε τέτοιου τομεί. Ευχαριστούμε κυρία Κοράτσα Μπίλτ. Ίσως θα χρειαζόμασταν εδώ ένα θερμόμετρο ε, ή ένα σφιγμομετρήσιμο να δούμε Ποιο είναι πολύ Ευρωπαίος, φιλοευρωπαίος, ποιο λιγότερο κτλ. Η κυρία Ιούτο έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια. Για μα. πραγματικά καταφέραμε να κάνουμε ως πολιτική ομάδα και ως αντιπροσωπεία μια πολύ καλή συνενετική επικοδομητική συνεργασία με την εισηγήτρια. Υποβάλαμε και εμείς κάποιες τροπολογίες και στα πλαίσια της Επιτροπής Απασχόλησης. Το ζήτημα αυτό μας απασχολεί ιδιαιτέρως. Σίγουρα λοιπόν υποβάλαμε κάποιες τροπολογίες που καλούν ε, την εναρμόνιση της νομοθεσίας από το ένα κράτος μέρος στο άλλο, προκειμένου να έχουμε μια ευρύτερη προστασία των κατηγοριών αυτών όσον αφορά την προστασία της υγείας των εργαζομένων, ή την επέκταση κάποιων δικαιωμάτων όπως το δικαίωμα μητρότητας και σχετικές υπηρεσίες. Εμείς στην Ιταλία έχουμε μια εθνική νομοθεσία, αλλά ξέρουμε ότι υπάρχουν και άλλα κράτη-μέλη στα οποία δεν υπάρχει τέτοια σχετική νομοθεσία προστασίας. Επομένως η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει σε κοινοτικό επίπεδο να ασχοληθεί με το ζήτημα αυτό, με την προστασία αυτών των κατηγοριών το θέμα δεν είναι αυτή τη στιγμή να δούμε πού έγκυται η αρμοδιότητα εθνική ή ενωσιακή. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να επεκτείνουμε ή να δημιουργήσουμε δικαιώματα εκεί πέρα που δεν υπάρχουν. Αν υπάρχουν κάποια κράτη-μέλη τα οποία δεν έχουν κάνει σπουδαία πράγματα, πρέπει να αναβαθμίσουν την νομοθεσία του. Υποβάλαμε τροπολογίε όσον αφορά την αύξηση των ελέγχων για τι επαγγελματικέ αυτέ κατηγορίε. Ξέρετε ότι πολύ συχνά δεν γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι και όταν γίνονται τελικά ενοχοποιούνται οι ίδιες οι εργαζόμενες. Είναι πολύ σημαντικό οι έλεγχοι αυτοί να λειτουργούν ως έλεγχοι προστασίας που θα υποβάλουν εχέγγυα για τις γυναίκες αυτές και όχι κυρώσεις ως προς αυτές. Πρέπει ουσιαστικά να προστατεύσουμε μέσω των ελέγχων το δικαίωμα στην εργασία. Νομίζω λοιπόν ότι και εκεί πέρα χρειαζόμαστε μια κάποια ευθυγράμμιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και υποβάλαμε και κάποιες άλλες τροπολογίες όσον αφορά την δημιουργία κάποιων επαγγελματικών προσόντων για τις οικιακές αυτές βοηθούς ή για το προσωπικό φροντίδας. Ξέρετε ότι πολύ συχνά οι γυναίκες αυτές πρέπει να ασχοληθούν είτε με παιδιά είτε με ιδιαίτερα ηλικιωμένους ανθρώπους. Δεν μπορούν λοιπόν να κάνει, να κάνει τη δουλειά αυτή οποιοδήποτε. Πολύ συχνά καταλαβαίνετε ότι επειδή οι θέσει αυτές απασχόλησης δεν πληρώνονται καλά, τελικά καλύπτονται από ανθρώπους που δεν έχουν τις απαραίτητες δεξιότητες. Αν κάποιος έχει συγκεκριμένε δεξιότητες, προφανώς δεν θέλει να υποπληρώνεται. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε ειδικευμένο προσωπικό, ανθρώπους με συγκεκριμένε δεξιότητες, οι οποίες θα μπορούν να πληρούν αυτές τις εργασίες και νομίζω ότι θα πρέπει βέβαια να έχουν και τις αντίστοιχες εξεπρεπείς ε, αποδοχές. Υποβάλαμε και μία ακόμα τροπολογία προκειμένου να δοθούν κάποια κίνητρα για την ε, έμεση παροχής ε, φροντίδας στο σπίτι. Ξέρετε ότι πολλές φορές άνθρωποι, για παράδειγμα, που πλήττονται από κάποια αναπηρία, μπορεί να επιλέγουν να έχουν στο σπίτι μια γυναίκα που θα μπορεί να τους βοηθήσει από το να πάνε σε κάποιο ειδικευμένο κέντρο υποδοχής και φροντίδας για την αναπηρία αυτή. Νομίζω λοιπόν ότι και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας και να προβλέψουμε στην έκθεση και συγκεκριμένες διατάξεις για το ζήτημα αυτό. Πάντως πέρα από τις μικρές αυτές διευκρινήσεις και τροπολογίες, θεωρούμε ότι το κείμενο είναι πολύ θετικό. Η κυρία Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Κούνεβε, ευχαριστώ πολύ. Εκτιμούμε πολύ την έκθεση και το περιεχόμενο. Ένα σχόλιο πρώτα απ' όλα σε σχέση με, το, με την αρμοδιότητα. Η υγεία και ασφάλεια στον χώρο εργασία είναι αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως μέλος της Επιτροπή ΕΜΠΛ, επίσης, περιμένουμε συνεχώ αυτού, διότι είναι ένα από τα πιο ισχυρά εργαλεία που έχουμε στα χέρια μας για να εξελίψουμε το dumping στην υγεία και την ασφάλεια στην εσωτερική αγορά. Ένα πραγματικό Ευρωπαίος πρέπει να δίνει μάχη υπέρ όλων αυτών, κυρία Κοράτσα Μπίλτ. Έχει μεγάλη σημασία επίσης να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν είναι μόνο το, η εργατική νομοθεσία. Εδώ έχουμε να κάνουμε με θεμελιώδη δικαιώματα των εργαζομένων, τα οποία πλήττονται από καταχρήσεις. Μιλάμε ύστερα για τράφικινγκ, για εμπόριο ανθρώπων και εδώ χρειαζόμαστε νομοθετική πρωτοβουλία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ακούστηκαν πολλά με τα οποία συμφωνώ κάτι πολύ σημαντικό για την ομάδα μου είναι το θέμα του τράφικινγκ και των εγκληματικών πρακτικών που συνήθως αντιμετωπίζουμε και αντιμετωπίζει ο χώρος των ε, εργαζομένων. Πολλές φορές η αστυνομία και οι δικαστές διαπιστώνουμε ότι χρειάζονται περισσότερη εκπαίδευση και κατάρτιση για να μπορούν ακριβώς να αντιμετωπίζουν ε, τις υποθέσεις αυτές προστατεύοντας τα δικαιώματα των εργαζομένων. Στην 11α τονίζεται αυτή ακριβώς η πτυχή. Ελπίζω ότι θα την υποστηρίξετε γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία, παραλαμβάνω, για την προστασία ιδιαίτερως των γυναικών αλλά και όλων των ανθρώπων που είναι του τράφικινγκ. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Κύριε Κότσα, θέλει να παρέμβει νομίζω. Ναι, ε, θα μιλήσω επί προσωπικού. Να διευκρινίσω κύριε Πρόεδρε, τι σημαίνει επικουρικότητα. Όταν λέω ότι είναι εθνική αρμοδιότητα, δεν σημαίνει ότι δεν μας νοιάζει, ότι δεν μας νοιάζει αυτή η κατηγορία εργαζομένων. Όχι, το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό, εννοείται. Αυτοί οι άνθρωποι δεν πρέπει να είναι αντικείμενα εκμετάλλευση. Πρέπει να την χάνουν αξιοπρεπού μεταχείριση και αντιμετώπιση όπως όλοι οι άλλοι εργαζόμενοι. Όμω η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι εδώ για να αντισταθμίζει τις παρελήψεις των κρατών Όχι, είναι εδώ για να παρέχει προσθεμένη αξία διασυνοριακά. Και θα συνεχίσω στα Ιταλικά, διότι θέλω να απαντήσω στην αγαπητή Σάλφα Ντανιέλα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να είναι μια ένωση η οποία θα καλύπτει τα κενά της εθνικής νομοθεσίας. Τα κράτη-μέλη είναι αυτά τα οποία πρέπει να πληρούν τις υποχρεώσεις τους, για παράδειγμα να καταπολεμήσουν την εκμετάλλευση των γυναικών αυτών, τους πάρα πολύ χαμηλούς μισθούς, το δεν υπάρχει νομοθετική κάλυψη. Δεν λέω ότι συμβαίνει αυτό στη Σουηδία, στην Ιταλία, αλλά συμβαίνει σε κάποια κράτη-μέλη. Όταν υπάρχουν τέτοια νομοθετικά κοινά, δεν μπορούμε εμεί να ερχόμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να λέμε ότι θα καλύψουμε τα νομοθετικά σα κενά, οτιδήποτε είπατε, η έλεγχη, το εργασιακό δίκαιο, το, το ότι οι γυναίκες αυτές πληρώνονται με πάρα πολύ χαμηλούς μισθούς, όλα αυτά είναι εθνικά καθαρά ζητήματα. Όλα αυτά τα ζητήματα δεν είναι διασυνοριακά, δεν μπορούν να διευθετηθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το ζήτημα το οποίο είναι διασυνοριακό είναι η εμπορία ανθρώπων. Έχουμε όμως μια οδηγία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εγώ είμαι η εισηγήτρια για την οδηγία εφαρμογή όσον αφορά την καταπολέμηση τη εμπορία ανθρώπων και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε τέτοια ευρωπαϊκή οδηγία για αυτό το ζήτημα όμω. Τώρα, όσον αφορά την εισηγήτρια. Το να νομοθετούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο κάθε φορά που προκύπτουν κενά σε εθνικό επίπεδο δεν νομίζω ότι είναι δικός μας ρόλος. Ο δικός μας ο ρόλος σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι να, να νομοθετούμε όταν μπορούμε να έχουμε μια προστιθέμενη αξία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μόνο τότε θα πρέπει να λαμβάνουμε δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και τώρα η κυρία Κυρία Πρόεδρε, πρώτον συγγνώμη για την καθυστερημένη μου άφηξη. Λοιπόν, για τις βεθούς; βυθού. Ε, ε, να σας πω και αυτό μια καλή είδηση. Στην Έμπλη μόλις υπερψηφίσαμε τη γνωμοδότηση υπέρ τη έκθεση, και καταφέραμε νομίζω να ενσωματώσουμε καλέ τροπολογίες οι οποίε θεωρώ ότι μπορούν να συμπεριληφθούν και στην έκθεση. Χαίρομαι διότι είχαμε καλά αποτελέσματα όπω είπα στην Apple να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, καταρχάς την κυρία Κούνεβα. Θεωρώ ότι θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε επί συγκεκριμένων τροπολογιών για να συντάξουμε μαζί συμβαστικές τροπολογίες. Και εγώ ως ε, έχω μερικές τροπολογίες. Και να μην υπησέλθω τώρα στις λεπτομέρειες. Θα τα δούμε αυτά. Λέω λοιπόν για άλλη μια φορά ότι προσβλέπω σε επικοδομητική συνεργασία. Πρόεδρος, πολύ ωραία για να κλείσουμε. Η κυρία Κούνεβα, νομίζω θέλετε το λόγο. Κυρία Κούνεβα ξανά. Ή κάνω λάθος. Σα ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις σας. Θα έχουμε την ευκαιρία να συνεργαστούμε και πιο στενά σε μια συνάντηση των σκιωδών εισηγητών. Όσον αφορά τους φόβους για τις νομοθετικές πρωτοβουλίες, θα ήθελα να τονίζω πως έχουμε κάθε δικαιώμα να προτείνουμε κατευθύνσεις ώστε να, τα κράτη-μέλη να αναλάβουν πρωτοβουλίες για καλύτερη προστασία. Δεν επεμβαίνουμε στο εθνικό δικαιό, προτείνουμε στα κράτη-μέλη με βάση τα δεδομένα που έχουμε για σοβαρά προβλήματα σε αυτόν τον τομέα να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να δράσουν τα κράτη-μέλη και η Κομισιόν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Ράινκε και την, για την παρατηρήση σε αυτήν την κατεύθυνση. Σε ευχαριστώ την κυρία Μπλίνκεβιτσιούτη, η οποία επιβιώσε πως μόλις ψηφίσαμε την Επιτροπή, την Επιτροπή Απασχόληση Μέτρα σε αυτήν την κατεύθυνση και θα ήθελα να κάνω ένα ερώτημα σε όλους μας εδώ, γιατί είμαι βέβαιη πως πολλοί από εμά χρησιμοποιούν οικιακά εργαζόμενος. Έχουμε αναρωτηθεί για τη ζωή αυτών των ανθρώπων. Σαν την αντιμετωπίζουμε σωστά, είναι εντελωμένοι, τους επιτρέπουμε να τηρούν τα νόμιμα ωράρια και τις σωστές συνθήκες εργασίας. Ευχαριστώ. Muchas eh, Σας ευχαριστούμε, κυρία Κούνεβα. Μετά από αυτή την ανταλλαγή απόψεων, θα προσέθετα μόνο το 17 Φεβρουαρίου, θα ξανασυζητήσουμε την έκθεση και μετά. Όχι, εγώ έκανα λάθος, ε, λέει η Πρόεδρος. Ζητώ συγγνώμη. 28 Ιανουαρίου θα γίνει η ψηφοφορία. Έχουμε χρόνο ε, για να ενσωματωθούν όλα τα σημεία μέσα στην έκθεση. Περνάμε στο επόμενο σημείο τώρα. Η ε, έκθεση της κυρίας Αρένα έχει μια προοπτική με γνώμονα το φύλλο. Ευχαριστώ η Ράτσε, θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Έστειλα στους σκιώδεις ένα έγγραφο εργασίας. Ε, θέλω να έχουμε πραγματικά χρόνο να επεξεργαστούμε την έκθεση και ήθελα να υπάρχει μια βάση εργασίας. Είπατε ότι έχουμε χρόνο για την προηγούμενη έκθεση και για τη δική μου, γιατί έχουμε προθεσμία μέχρι τον Ιανουάριο και ψηφίζουμε τον Απρίλη. Δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Τρεις είναι οι άξονες ε, ε στους οποίους θα βασιστούμε. Πρώτον, διαπίστωση σε σχέση με την συνεκτίμηση της διάθεσης του φύλου για το θέμα της φτώχειας με τη στρατηγική 2020 που στόχο είχε να μειώσει τη, γενικότερα τη φτώχεια στην Ευρώπη, όχι μόνο σε σχέση με το φύλλο. Τέλος, ε, όμως, ε, με την κρίση δεν υλοποιήθηκαν αυτοί οι στόχοι. Το αντίθετο, είδαμε ότι σε σχέση με τη φτώχεια έχει επιδεινωθεί η κατάσταση ως προς την, ε, τα δικαιώματα των δύο φύλων. Πλήττονται περισσότερο οι γυναίκε από τη φτώχεια λοιπόν ε, και επιδεινώνεται η κατάσταση. Δεύτερον, πέρα από το υλικό κομμάτι υπάρχει και το θέμα της στέρησης ε, ως προς την πρόσβαση ε, στον πολιτισμό, αποκλεισμός της γυναίκας από διάφορους τομείς της κοινωνίας λοιπόν πέρα από το υλικό κομμάτι πρέπει να δούμε σφαιρικότερα το ζήτημα. Τρίτον, ε, οι αιτίε τη φτώχεια. Φυσικά θα επανέλθουμε στο μισθολογικό χάσμα. Υπάρχουν και φτωχοί σε εισαγωγικά τομείς όπου επικρατούν οι γυναίκες. Τα είπαμε και νωρίτερα ε, για τις οικιακές βοηθούς Εκεί ε, είναι έντονο το φαινόμενο της φτώχειας και με συντριπτική πλειοψηφία των γυναικών. Ε, οι οικογενειακές δομές επίσης, αν δεν ληφθούν όντως υπόψη, μπορεί να ε, οδηγήσουν σε μεγαλύτερη φτώχεια. Επίσης υπάρχει το θέμα του χάσματος ως προς τη συντάξη, δηλαδή για τις ηλικιωμένες γυναίκες, Βλέπουμε λοιπόν ένα συνδυασμό ε, διαφόρων ε, τομέων όπου παρατηρείται το φαινόμενο της στόχιας. Δεύτερο κομμάτι, οι λύσεις. Πρώτον, ενεργοποίηση νομοθετικού χαρακτήρα. Τι εννοώ, ποια είναι τα μέτρα που λειτουργούν αισίως, ποια όχι και ποιες τροποποίησεις μπορούμε να επιφέρουμε στα νομοθετικά μέσα. Δεύτερον, μέτρα ε, με προσαρμογή των κονδυλίων στον προϋπολογισμό. Με ποιο τρόπο μπορούμε να καταπολεμήσουμε τη φτώχεια με ε, μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας ε, εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τον προϋπολογισμό και πώς μπορούν να υλοποιηθούν. Τρίτον, ανταλλαγή βελτίστων πρακτικών όταν βλέπουμε για το φορολογικό ζήτημα και συμφωνώ με την ε, κυρία Κοράτσα Μπίλτη υπάρχουν ε, εθνικές αρμοδιότητες όπως η φορολογία. Υπάρχουν ε, όμως και παράγοντες που δημιουργούν, εντείνουν, οξύνουν το φαινόμενο της φτώχειας σε επίπεδο ε, κράτους μέλους και θα πρέπει λοιπόν να διαπιστωθούν ποιοι είναι αυτοί οι παράγοντες και να ε, γίνει και ανταλλαγή πρακτικών. Αυτή είναι η τρεις βασικοί άξονες. Έχουμε ήδη συνεργαστεί με τους σκιώδεις και περιμένω τα σχόλιά τους, ούτω ώστε να έχουμε ήδη ένα ε, συνενετικό κείμενο για να συνεργαστούμε περαιτέρω. Σας ευχαριστούμε κυρία Ρένα. Τώρα περνάμε στις ε, ε συναδέλφους. Τσούμπερ. Συγγνώμη, κυρία Σουίτσα και όχι κυρία Τσούμπερ. Θα ήθελα ως σκιώδης εισηγήτρια πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την κυρία Ρένα για το έγγραφο εργασίας. Βρίσκονται η κατανομή αυτά τα τρία τμήματα, στις τρεις άξονες είναι καλή. Κάναμε μια σύντομη ανταλλαγή απόψεων. Εγώ νομίζω ο βασικός στόχος πρέπει να είναι η καταπολέμηση της φτώχειας. Ε, μιλήσαμε και για την ε, οικονομική κρίση, ότι δεν υλοποιήθηκαν οι στόχοι ε, που είχαμε προσδιορίσει. Θα πρέπει λοιπόν να ξέρουμε ακριβώς ποιες ήταν οι επιπτώσεις στις γυναίκες και πώς μπορούν να ξεφύγουν από αυτή την κατάσταση, διότι δεν είναι μόνο υλικό το ζήτημα, όπως είπε και η κυρία Ρένα, είναι και θέμα υπηρεσιών, αλλά φυσικά μπορούμε από οικονομικής πλευράς να εξετάσουμε το θέμα της πρόσβασης, της καθολικής πρόσβασης στις υπηρεσίες εξετάζοντας ε, την κατάσταση και κάνοντας ε, τις συγκρίσεις ανάμεσα σε αναπτυσσόμενες και αναπτυγμένες χώρες διαπιστώνουμε ότι είναι παρεμφερή δυστυχώς τα προβλήματα, χρειάζεται αλλαγή ε, και κυρία Ρένα μιλήσατε και για νομοθετική παρέμβαση. Εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι και το σημαντικότερο ζήτημα το ζήτημα της μετρικής άδειας, το ζήτημα της επικουρικότητας, τι μπορούμε να, αποφύγουμε, να αποφασίσουμε συγγνώμη, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και τι μπορούμε να ε, ρυθμίσουμε σε επίπεδο κράτους μέλους. Φυσικά ε, υπάρχει το φορολογικό ζήτημα, ζήτημα εθνικής αρμοδιότητας, ε, το ξέρω αυτό, είναι εθνικό ζήτημα όμως παρόλα αυτά γίνεται μέσα σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε άλλες επιτροπές για τη φορολογία και το θέμα ποιο είναι να υπάρχει ίση φορολόγηση ώστε να υπάρχει ε, και μεγαλύτερη συνοχή. Ε, για η ίση αμοιβή παραδείγματος χάρη για την ίδια εργασία. Νομίζω ότι είναι εκ των κάνευ ε, προϋπόθεση για να μπορέσουμε να σημειώσουμε πρόοδο. Ελπίζω λοιπόν να συνεχίσουμε αυτή την ε, πολύ καλή συνεργασία που έχουμε και να τελείξουμε σε ένα συνεργατικό κείμενο. για να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε αυτήν την εκμετάλλευση του ε, αδυνάμου φίλου που θα ήθελα τώρα να δώσω, λέει το λόγο η πρόεδρος, στην κυρία Βυσνιεύσκα και το προφέρω και πάλι σωστά το όνομά σας. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Αναμφίβολα οι γυναίκες εκτίθενται περισσότερο στη φτώχεια. Και το γεγονός ότι οι γυναίκες βέβαια είναι και μητέρες. Αυτό δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο την θέση στην οποία βρίσκονται. Επίσης λαμβάνουν, όπως είπε και η συγγήτρια, χαμηλότερους μισθούς και στη συνέχεια χαμηλότερες συντάξεις. Επίσης αυξάνονται όλο και περισσότερο τα διαζύγια και το αποτέλεσμα είναι ότι οι μονογονεϊκές οικογένειες που έχουν αρχηγό γυναίκα βρίσκονται σε όλο και πιο δεινή θέση Πρέπει λοιπόν να, να ληφθεί δράση προκειμένου να μικρύνει το μισθολογικό χάσμα και να καταφέρουμε να συμφιλιώσουμε καλύτερα επαγγελματική και προσωπική ζωή. Όσον αφορά τώρα το επίπεδο των μισθών, δεν υπάρχει καμία απολύτως δικαιολογία για να έχουμε διαφορετικούς μισθούς μεταξύ ανδρών και γυναικών για την ίδια θέση απασχόλησης. Δυστυχώς όμως αυτό συμβαίνει στην πράξη. Ας μην έχουμε λοιπόν ε, ψευδεστήσεις. Το χάσμα αυτό δεν πρόκειται να εξαλειφθεί εντελώς. Γι' αυτό ακριβώς τουλάχιστον για να είμαστε πιο ρεαλιστές θα πρέπει να λέμε ότι θέλουμε να περιορίσουμε το μεσολογικό χάσμα και όχι να το εξαλείψουμε. Νομίζω ότι θα σημειώσουμε επιτυχία να αρχίσουμε καταρχάς μειώνοντας το μεσολογικό αυτό χάσμα. Μπορεί να υφίσταται το χάσμα αυτό διότι ε, οι άντρες τελικά καταλαμβάνουν πιο διευθυν, περισσότερες διευθυντικές θέσεις ε, στις επιχειρήσεις. Η δική μου πολιτική ομάδα, το ECR, δεν θέλει δεσμευτικές ποσοστώσεις για τις γυναίκες σε καμία περίπτωση. Όχι διότι θεωρεί ότι οι γυναίκες είναι κατώτερες, αλλά διότι οι γυναίκες πολλές φορές ε, επιτελούν και διαφορετικούς κοινωνικούς ρόλους οι γυναίκες με το να ασχολούνται με τα παιδιά ενδεχομένω να μην έχουν τον απαραίτητο χρόνο για να ασχοληθούν με την επαγγελματική τους καριέρα. Και αυτό πρέπει να το αναφέρουμε και να τονίσουμε το ρόλο της γυναίκας στην κοινωνία ως μητέρα. Νομίζω λοιπόν θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλες τις ε, μεθόδους που έχουμε στη θέση μας προκειμένου να συμφιλιώσουμε επαγγελματική και προσωπική ζωή. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε πιο ευέλικτες μορφές άδειας μητρότητας, προκειμένου οι γυναίκες να μπορούν να επιστρέφουν πιο μαλά και πιο αποτελεσματικά στην αγορά εργασίας. Ως προς αυτό δεν νομίζω ότι έχουμε καμία αμφιβολία, από καμία πολιτική ομάδα θα υπήρχε κάποια αντίρρηση. Ωστόσο, θα πρέπει να έχουμε κατά νου και το ζήτημα των συντάξεων. Οι γυναίκες οι οποίες εγκατέλειψαν την επαγγελματική ζωή προκειμένου να ασχοληθούν με την ανατροφή των παιδιών τους. Γίνεται μια αναφορά λοιπόν στην περίπτωση αυτή και γίνεται μια αναφορά επίση στις γυναίκες αυτές οι οποίες εργάζονται σε παιδικούς σταθμούς και ουσιαστικά λαμβάνουν μισθό για την εργασία που επιτελούν άλλες γυναίκες μένοντας στο σπίτι τους. Γίνεται περαιτέρω επίσης μία αναφορά στις φορολογικές υποχρεώσεις των γυναικών και εκεί πέρα νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει μια ισότιμη αντιμετώπιση σε σχέση με τους άντρες. Έχω λοιπόν να κάνω τρεις συγκεκριμένε ερωτήσεις προς την εισηγήτρια. Τι εννοείτε όταν λέτε ότι θα πρέπει να υπάρχουν ε, εξατομικευμένα δικαιώματα στα πλαίσια των οικοκυριών όσον αφορά τις φορολογικές υποχρεώσεις. Δηλαδή, εκ των προτέρων και αναλογικά θα πρέπει να έχουμε φορολογικές υποχρεώσεις με βάση το μισθό που λαμβάνει το κάθε μέλος ενός νοικοκυριού. Και μία ακόμα ερώτηση. Πώς μπορούμε να έχουμε μία ισότιμη συμβολή και των ανδρών στα οικιακά, στις γενικότερες υποχρεώσεις οι οποίες προκύπτουν στα πλαίσια ενός νοικοκυριού. Πώς μπορεί να επιτευχθεί κάτι τέτοιο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Νομίζω ότι προφέρετε καλύτερα το δικό μου το επίθετο, έτσι δεν είναι. Να ευχαριστήσω την κυρία Ρένα για αυτό το έγγραφο εργασία το οποίο υπέβαλε. Είναι το πρώτο βήμα προτού εμπλακούμε περισσότερο με τη σύνταξη της έκθεσης, την κατάθεση τροπολογιών και την οριστικοποίηση του τελικού εγγράφου. Έχοντας όντως ένα έγγραφο εργασία ήδη από τώρα στα χέρια μας, μπορούμε και εμείς να αρχίσουμε μία ώρα αρχίτερα την εργασία που πρέπει να κάνουμε. Θεωρώ ότι είναι πολύ θετικό το ότι αναφέρεται το ότι δεν βλέπουμε την φτώχεια των γυναικών. Είναι πολλές φορές αόρατη, δεν την παρατηρούμε καθόλου. Κανείς δεν ασχολείται με αυτή την κατηγορία ένδυας. Το γεγονό ότι δεν βλέπουμε πάρα πολλέ γυναίκε να ζητιανεύουν στου δρόμου δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν αρκετέ φτωχέ γυναίκε στις κοινωνίες μα. Τα βασικότερα σημεία της έκθεσης αυτής θεωρώ ότι είναι καταρχάς το μισθολογικό χάσμα, το ότι πολύ συχνά έχουμε γυναίκες οι οποίες αναλαμβάνουν την ανατροφή των παιδιών ότι πολλές φορές γυναίκες σε μονογονεϊκές οικογένειες όχι μόνο έχουν χαμηλούς μισθούς στην αρχή, αλλά καταλήγουν και με πενιχρές συντάξεις. Επίσης εστιάζεστε, κυρία Ρένα, πολύ στις μονογονεϊκές οικογένειες και όντως ένα 85% των οικογενειών αυτών έχουν γυναίκες ως αρχηγούς. Το ζήτημα αυτό το έχουμε αναλύσει και στην χώρα μου, την Ισπανία, και είναι γενικότερα η δεδομένη εικόνα αυτή των μονογονεακών οικογενειών που ουσιαστικά παρτίζονται από μία γυναίκα και ένα ή περισσότερα παιδιά. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να ασχοληθούμε ακριβώς με αυτή την κοινωνική κατηγορία πλέον. Σπάνια βλέπουμε μονογονεακές οικογένειες που παρτίζονται κυρίως από έναν πατέρα και παιδιά. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε πολύ με αυτή την κατηγορία. Είναι επίση πάρα πολύ θετικό το ότι ε, η συγγήτρια αναφέρεται στη γενικότερη απογοήτευση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όταν ενημερώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι πρόκειται να αποσύρει την πρόταση νομοθεσία για την άδεια μητρότητα. Νομίζω ότι πρέπει να ασχοληθούμε επίση και με το ζήτημα τη φροντίδα των ε, παιδιών. Όπω είπαμε πολλέ φορέ, μόνε γυναίκε αναγκάζονται να ασχοληθούν με το ζήτημα αυτό χωρί να έχουν καμία απολύτω υποστήριξη. Νομίζουμε ότι μεγαλύτερη έμφαση επίσης θα πρέπει να δοθεί στον αντίκτυπο των γενικότερων πολιτικών λιτότητος. Λέγεται αυτό ήδη στο κείμενό σας, γίνεται μια σύντομη μνήμα, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να το προβάλλουμε ακόμα περισσότερο. Έχουν μειωθεί οι δημόσιες υπηρεσίες, έχουν μειωθεί οι παιδικοί σταθμοί και πάρα πολλές γυναίκες σε ορισμένες χώρες αναγκάστηκαν να σταματήσουν να εργάζονται μόνο και μόνο για να ασχοληθούν με τα παιδιά τους, ακριβώς επειδή το κράτος δεν είναι πλέον σε θέση να παράσχει αυτές τις πολύ βασικές υπηρεσίες φροντίδας των παιδιών. Νομίζω επίσης ότι θα πρέπει να δούμε και πώς έχει η εξωτερική μας πολιτική, η πολιτική οικονομική ανάπτυξης, στην οποία προωθούμε προς τρίτες χώρες. Δεν νομίζω ότι στην πολιτική συνεργασία που έχουμε, στι εμπορικέ συμφωνίε που συνάπτουμε με τρίτε χώρε, δεν κάνουμε αρκετή αναφορά στην ε, μείωση τη φτώχεια όσον αφορά τι γυναίκε ή στην πρόθεση τη ισότητα των φύλων. Νομίζω ότι οι δύο συναπτυσσόμενε χώρε θα πρέπει να ασχοληθούμε πάρα πολύ με αυτό το ζήτημα τη εξάλληψη τη γυναικεία φτώχεια. Η δική μου επίση πολιτική ομάδα θα ήθελε να γίνεται σαφή αναφορά στην προθεση τη ισοτητα των θυλων νομιζω οτι οι δυο συναπτυσσομενε χωρε θα πρεπει να ασχοληθουμε παρα πολυ με αυτο το ζητημα τη εξαλληψη τη γυναικεια φτωχεια η δικη μου επιση πολιτικη ομαδα θα ηθελε να γινεται σαφη αναφορα στην εκθεση σα στην λεγόμενη κλιματική δικαιοσύνη και αναφέρομαι επίσης και στις όλες τις συζητήσεις που λαμβάνουν αυτή τη στιγμή χώρα στο Παρίσι. Ξέρετε ότι είναι οι γυναίκες αυτές οι οποίες πλήττονται κυρίως από τις κλιματικές αλλαγές. Πρέπει να προστατεύσουμε και τις γυναίκες αυτές και θα πρέπει να καταφέρουμε να δούμε πώς μπορούμε να θεραπεύσουμε όλες αυτές τις αρνητικές επιπτώσεις. Και μία τελευταία παρατήρηση. Γνωρίζω ότι δεν υπάρχει ευρύτερη υποστήριξη για το ζήτημα αυτό, ωστόσο θα θέλαμε να γίνεται μια κάποια αναφορά σε ένα βασικό ελάχιστο μισθό προκειμένου να μπορούμε τουλάχιστον να αντιμετωπίσουμε εν μέρη το πρόβλημα αυτό της φτώχειας που πλήττει τις γυναίκες. Έναν καθολικό ελάχιστο μισθό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω την συγκήτρια που υπέβαλε αυτό το αρχικό έγγραφο εργασία. Θεωρούμε ότι είναι πολύ θετική η διαδικασία που ακολουθεί και πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε μια πολύ θετική έκθεση. Σας ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομη. Ε, η κυρία Ζήπερνε είναι ισχυώδης μας, αλλά δεν μπορούσε να έρθει, να, να μείνει μάλλον στη συνεδρίαση. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτό το έγγραφο εργασίας όπως το ονομάζεται, που είναι μια κοινή άποψη για τα σημαντικότερα ζητήματα που θέλουμε να θέσουμε. Λέγουμε τι αιτίε λοιπόν τη φτώχεια και αυτό είναι κάτι που πρέπει να τονίσουμε και όπως ε, είπαν ε, και οι συνάδελφοι θα πρέπει να μιλήσουμε για την κρίση και τις επιπτώσεις που είχε. Να τονίσουμε ότι υπάρχουν ομάδες που πλήττονται περισσότερο από τη διακριτική μεταχείριση μονογονιακής οικογένειας, ηλικιωμένες ε, γυναίκες και το χρειαζόμαστε ε, ιδιαίτερες πολιτικές για να καταφέρουμε να καταπολεμήσουμε τη φτώχεια σε αυτές τις ε, πληθυσμιακές ομάδες, ε, η φροντίδα των παιδιών, το θέμα της γονικής και μητρικής άδειας και συμφιλίωση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής είναι ζητήματα που πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να φέρουμε βελτιώσεις είτε σε ενωσιακό επίπεδο είτε σε εθνικό επίπεδο όπου πρόκειται για θέματα ε, ε, κορικότητας. Χρειάζεται να εξασφαλίσουμε ε, την οικονομική ανεξαρτησία και τα κοινωνικά ασφαλιστικά συστήματα για τις γυναίκες για να μπορούμε να επιτύχουμε την αυτοδιάθεση των γυναικών. Αυτό διαπιστώνουμε από την εμπειρία μας στη Σουηδία. Ήδη στην δεκαετία του 70 ασφαλίζονταν προσωπικά οι γυναίκες και όχι σε σχέση με τους συζύγους τους ε, και αυτό οδηγεί σε μεγαλύτερη ανεξαρτησία και είχε τα πάρα πολύ θετικά αποτελέσματα που γνωρίζουμε στη Σουηδία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κυρία Μπιόρκ. Ευχαριστώ. Καταρχάς, συγγνώμη για την καθυστέρηση. Έπρεπε να είμαι σε άλλη συνεδρίαση για ένα κακό υπολογισμό χρόνου. Πάση περιπτώσει, εδώ ελπίζω να ακούσω την ισχύτρια. Για το κείμενο καταρχήν. Συγχαρητήρια για το έργο που έγινε τώρα. Η ισχύτρια έκανε σπουδαία δουλειά. Πρέπει όμως όλα αυτά να τα συνοδεύσουμε και με άλλε πρωτοβουλίε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Να υπάρχει στοιχειώδης αυτοσυνέπεια θα λέω ότι πρέπει να τονίσουμε περισσότερο δύο πράγματα. Πρώτον, να συνειδητοποιήσουμε ότι η φτώχεια των γυναικών σε πολλές περιπτώσεις εξαρτάται, συναρτάται με την έλλειψη προσόντων ή εκπαίδευσης και κατάρτισης. Με άλλα λόγια, αυτές οι γυναίκες οθούνται ουσιαστικά προς ε, χειρότερα πληρωμένες δουλειές εκ των πραγμάτων. Άρα το ζητούμενο είναι εκπαίδευση και κατάρτιση. Να συνειδητοποιήσουμε την αιτία του προβλήματος. Να βοηθήσουμε τις γυναίκες να συμμετάσχουν σε, σε προγράμματα ε, της τοπικής αυτοδιοίκησης ή και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να παρακολουθούν μαθήματα πάνω σε επιστημονικούς τομείς, τεχνικούς τομείς. Επίσης η επαγγελματική κατάρτιση είναι πολύ σημαντική προκειμένου. Το βλέπουμε ότι το λεγόμενο μεικτό σύστημα τη ε, επαγγελματική κατάρτιση είχε αποτελέσματα. Βελτιώνουμε δηλαδή την απασχολησιμότητα των γυναικών. Το δείχνουν και τα στοιχεία. Δυστυχώ, ε, οι γυναίκε δεν συμμετέχουν αρκετά σε αυτέ τι πρωτοβουλίε δεν είναι αρκετά ενημερωμένες. Να τις ενημερώσουμε. Η εκθεσή τους ε, σε μαθήματα και τεχνολογίας σίγουρα θα τις βοηθήσει. Θα λέγατε είναι το κλειδί. Δεύτερον, ε, δεν ξέρω αν κατάλαβα καλά, αλλά στην έκθεση διατυπώνεται ότι υπάρχει σχέση μεταξύ φτώχειας και κακομεταχείρισης και καταχρήσεων εις των γυναικών. Δεν ξέρω, υπάρχουν όντως στοιχεία περί αυτού. Εδώ ξέρουμε ότι υψηλά ιστάμενα στελέχη, γυναίκες, ε, μορφωμένες ε, σε μεγάλες επιχειρήσεις και αυτές εκτίθενται σε παρενόχληση, πιέση κλπ. Δεν ξέρω αν υπάρχει λοιπόν αναγκαστικά συσχετισμός μεταξύ ε, κακομεταχείρισης, πιέσεων κλπ. παρενόχλησης και φτώχειας. Σε κάθε περίπτωση οφείλουμε να βγάλουμε τις γυναίκες από τη φτώχεια. Να τους εγγυηθούμε αν είναι δυνατόν, ένα ελάχιστο εγκυμένο εισόδημα. Να δημιουργήσουμε ένα εργαλείο ώστε να μπορούμε να του εγγυηθούμε ένα ελάχιστο κειμένο εισόδημα στην Ευρώπη. Γιατί, διότι όπου αυτό είναι πραγματικότητα, πέτυχε στην χώρα των Βάσκων και ενάντια σε τεράστια αντίδραση τώρα είχαμε κρίση, ανεργία εισηχθεί το εγκείμενο εισόδημα το οποίο βοήθησε ανθρώπους σε ακραία ένδια να προχωρήσουν και να επανενταχθούν. Λοιπόν, πέρασαν από τώρα 25 χρόνια. Σήμερα έχουμε μια πιο συνεκτική κοινωνία και έχουμε μάθει το μάθημά μας. Ιδιαίτερα ε, δεδομένη στις σοβούσα κρίση, κάτι παρόμοιο πρέπει να κάνουμε. Γιατί ο κόσμο θέλει να δουλέψει. Γιατί δουλειά σημαίνει αξιοπρέπεια. Να δημιουργήσουμε λοιπόν αποτελεσματικά εργαλεία για να του βοηθήσουμε. Υπάρχει σχετική εμπειρία. Και νομίζω ότι αν το κάνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τόσο το καλύτερο. Αυτέ είναι οι προτάσει μου, πέραν των ε, προτάσεων βεβαίω που περιέχει το κείμενο. Και τέλο, να πούμε και δύο λόγια για τι γυναίκε με αναπηρίε. Οι γυναίκε με αναπηρίε αντιμετωπίζουν ακόμη πιο σύνθερα προβλήματα ω προ την φτώχεια. Είναι γυναίκε, υποφέρουν από αναπηρίε, ε, έχουν άλλε δυσκολίε, μπορεί να έχουν και παιδιά. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πρέπει να προβάλλουμε και αυτό το πρόβλημα εδώ στο Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Πάω στο κύριο Βιλπάου. Κυρία Αρένα. Ευχαριστώ. Για όλες τις ε, ιδέες που κατατέθηκαν, πήρα σημειώσεις. Βλέπω, καταλαβαίνω πώς μπορούμε να συμπληρώσουμε το κείμενο, να το βελτιώσουμε. Προκύπτει ένα θέμα με πιο εντερό τρόπο. Ιδιαίτερος προς την έννοια του ατομικού φορολογικού δικαιώματος, της, ατομικής, της εξατομικευμένης φορολογικής μεταχείρισης, αν θέλετε. Δηλαδή, στις περισσότερες περιπτώσεις, η κοινή δήλωση είναι εις βάρος της γυναίκας σε ένα νοικοκυριό. Εμείς θέλουμε, ανεξαρτήτως αυτού, φορολογική μεταχείριση να είναι εξατομικευμένη. Να μην σωρεύεται δηλαδή το εισόδημα μια γυναίκα με αυτό του συζύγου. Αυτό θέλουμε. Πλήρη εξατομικευσή. Όπω το είπε και η Μπιόρκ. Αυτό προϋποθέτει και εξατομικευμένη μεταχείριση σε επίπεδο κοινωνικής ασφάλισης εν γέννη και βεβαίω δικαιωμάτων εν γέννη. Είμαι γυναίκα, δεν θέλω να θεωρούμε ως προσάρτημα κάποιου άνδρα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τους σκοπούς της φτώχειας. Κατά τα άλλα κρατέθηκαν πολλές ενδιαφέρουσες ιδέες. Πρέπει να εμπνευστούμε και από άλλες εκθέσεις. Σύμφωνοι για τις ε, γυναίκες με αναπηρίες μάλιστα έχουν υποθεί πολλά άλλα πράγματα. Θα διαβάσω τις σχετικές εκθέσεις και η Julie Ward το είπε. Μίλησε επίσης για τις αγρότησες που αντιμετωπίζουν σε ορισμένε περιπτώσει ε, εξαιρετικά δύσκολε συνθήκε, όπω όλοι οι αγρότε, βέβαια γενικότερα. Ναι, θα προσθέσω πολλά πράγματα. Φυσικά δεν μπορούμε να κάνουμε μια τεράστια έκθεση με 50 σελίδε. Θα προσπαθήσω να τα συνθέσω όλα αυτά με το πιο οικονομικό για το κείμενο τρόπο. Πρόεδρο, ευχαριστώ πολύ, κυρία Ρένα. Ακόμη δεν έχουμε καταλήξει το χρονοδιάγραμμα. Αλλά όπως γνωρίζετε θα έχουμε μια πρώτη συζήτηση και θα δούμε μετά θα οριστικοποιήσουμε το χρονοδιάγραμμα για τις ψηφορίες και το καθεξής. Και τώρα θα με εργαστεί λίγο κύριε Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη και για αυτή την καθυστέρηση. Λοιπόν, το επόμενο σημείο στη μερίσια διάταξη έχει να κάνει με τη βιομηχανία νυφών κατά παραγγελία. Ο κλάδος αυτός στην Ευρώπη είναι νόμιμος, παρουσιάζει ανάπτυξη, αλλά δεν υπάρχουν συγκεκριμένες ρυθμίσεις. Τα γραφεία αυτά συνοικισεών λοιπόν λειτουργούν νόμιμα, αλλά βλέπουμε ότι ε, ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν καθιστά τις γυναίκες όλο και πιο ευάλωτες. Οι γυναίκες είναι αντικείμενο πολλές φορές κακομεταχείρισης, εκμετάλλευσης, απομόνωσης με την κυρία Χόνιμπολ και την κυρία Ρένα ήδη από το Μάρτιο. Το Μάρτιο του 2015 υποβάλαμε σχετικό ερώτημα. Όσον αφορά τη βιομηχανία νηφών κατά παραγγελία, είχαμε και μια εκδήλωση εδώ πέρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είμαστε πάρα πολύ απογοητευμένε με το χρόνο που χρειάστηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μα απαντήσει. Απάντησε μόνο τον Οκτώβριο η Επιτροπή και μάλιστα δεν απάντησαν καν στι ερωτήσει μα. Γι' αυτό το λόγο ζητήσαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποστείλει εδώ στην Επιτροπή μα μία εκπρόσωπο, προκειμένου μη τι άλλο να γίνει μαζί τη μία ανταλλαγή απόψεων για αυτό το ζήτημα. Θα ήθελα λοιπόν να καλέσω την εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την κυρία Άννα Εξτέντ, από το γραφείο του συντονιστή τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την καταπολέμηση τη εμπορία ανθρώπων, να μα κάνει μία παρουσίαση και αν μη τι άλλο να μα δώσει κάποιε καλύτερε και πιο επαρκεί απαντήσει στα ερωτήματά μα. Σα δίνω λοιπόν το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Όντω εκπροσωπώ το γραφείο του Συντονιστή τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την καταπολέμηση τη εμπορία ανθρώπων. Σα ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση αυτή. Κύριε Βασιλιάδου, δεν μπορούσε να τον παρούσα. Αναφερόμαστε εδώ πέρα σε μια νέα οδηγία καταπολέμηση εμπορία ανθρώπων. Είναι μια φιλόδοξη πρόταση που ατενίζει το μέλλον, υποστηρίζει τα ανθρώπινα και θεμελιώδη δικαιώματα, μια νομοθεσία που επικεντρώνεται στα παιδιά, στα θύματα και βασίζεται βέβαια και στη διάσταση του φύλου. Οι περισσότερες, όχι όλες, από τις νύφες αυτές κατά παραγγελία είναι πολλές φορές θύμα οικογενειακής βίας ή καταγκαναστικού γάμου. Αυτό παραβιάζει προφανώς τα θεμελιώδη δικαιώματά τους και βέβαια συμβάλλει σε μία ανισότητα με βάση το φύλλο. Η οδηγία λοιπόν για την προάσπιση των θυμάτων αυτών προβλέπει συγκεκριμένα δικαιώματα για την προάσπιση των θυμάτων και των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, εκεί πέρα εντοπίζονται ως ιδιαίτερα ευάλωτες ομάδες τα θύματα αυτά. Προβλέπονται λοιπόν ότι θα υπάρχει μια συγκεκριμένη προστασία από τον εκφοβισμό και επίσης το ένταλμα προστασία τη Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπει τη δυνατότητα προστασία των ανθρώπων αυτών όταν ταξιδεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το καθεστώς προστασίας δεν θα πρέπει να βασίζεται καθόλου στην χώρα καταγωγή, στη χώρα διαμονής των θυμάτων αυτών. Είναι πολύ σημαντικό σε κάθε περίπτωση ενδοκογενειακής βίας, κακομεταχείρισης κτλ. το θύμα και συγκεκριμένα η γυναίκα να μπορεί να έχει την απαραίτητη προστασία. Δεν είναι βέβαια όλες οι νύφες κατά παραγγελία θύματα εμπορίας ανθρώπων, ορισμένος όμως είναι και για τις περιπτώσεις αυτές ισχύει η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Έχουμε κυρίως βέβαια γυναίκες ή πολλές φορές νέες κοπέλες οι οποίες είναι θύματα εμπορίας ανθρώπων, θύματα καταναγκαστικής, καταναγκαστικών γάμων ή συνοικεσίων στα οποία βέβαια δεν έχουν δώσει τη σύμφωνη γνώμη τους. Ξέρετε εδώ πέρα ότι οι έννοιες αυτές αντιμετωπίζονται ξεχωριστά από νομικής πλευράς. Θέλοντα λοιπόν να αντιμετωπίσουμε το οργανωμένο έγκλημα και έχοντα το συγκεκριμένο πρόγραμμα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θέλουμε να καταπολεμήσουμε όλε αυτέ τι μορφέ εμπορία ανθρώπων ή καταναγκαστικών γάμων. Θέλουμε επίση να στεστούμε κυρίω ε, ε, στο ρόλο που μπορούν να δραματίσουν οι προξενικέ αρχέ καθώ επίση και οι συνοριοφυλακέ. Θεωρούμε ότι τρίτες χώρες είναι πάρα πολύ σημαντικό να αναλάβουν δράση και οι πρεσβείες και οι προξενικές αρχές για να αποφευχθούν τέτοια φαινόμενα. Η βιομηχανία νηφών κατά παραγγελία μπορεί να ενταχθεί στο γενικότερο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πρόληψη της εμπορίας ανθρώπων. Είναι σαφές ότι χρειάζεται να υιοθετήσουμε συγκεκριμένα μοντέλα προληπτικά προκειμένου να καταφέρουμε να μειώσουμε τα φαινόμενα αυτά και να υποστηρίξουμε τις πιο ευάλωτες ομάδες. Η όλη αυτή συζήτηση σχετίζεται επίσης και με τα συνοικέσια και τους καταναγκαστικούς γάμους. Πολλές φορές οι όροι αυτοί δεν είναι σαφείς, πολλές φορές υπάρχει μια σύγχυση ανάμεσα στο καταναστικό γάμο, το συνοικέσιο ή άλλες μορφές καταναγκαστικών γάμων. Για τις περιπτώσεις αυτές δυστυχώς σε πολλά κρατημέλη δεν υπάρχει σχετική νομοθεσία. Επίσης στο πλαίσιο νομοθεσίας Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εμπορία των ανθρώπων δεν γίνεται σχετική μνήμα. Κάθε φορά που ο καταναγκαστικός γάμος σχετίζεται με το φαινόμενο της εμπορίας ανθρώπων, μιλάμε για θύματα εκμετάλλευσης, κακομεταχείρισης. Πολύ συχνά έχουμε γυναίκες οι οποίες ε, ουσιαστικά πολλούνται μέσω συγκεκριμένων ιστοσελίδων. Πολύ συχνά Πρόκειται για γυναίκε από τρίτες χώρες οι οποίες επιθυμούν να έρθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μέσω του γάμου να καταφέρουν να εξασφαλίσουν μόνιμη διαμονή εδώ. πολλές φορές ε, δεν ε, μένουν σε μία χώρα, αλλά μετακινούνται από τη μία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην άλλη και πολλές φορές στη μετακίνηση αυτή πέφτουν θύματα διαφόρων ομάδων διακίνησης, παράνομης διακίνησης ανθρώπων. Έχει ασχοληθεί με το ζήτημα αυτό η Europol. Κατά τη διάρκεια της Λετωνικής επίσης Προεδρίας ασχοληθήκαμε με το ζήτημα αυτό. Η ε, Λετωνία έθιξε το ζήτημα αυτό πολύ έντονα κατά τη διάρκεια της δικής της Προεδρίας. Εμπορία και εκμετάλλευση γυναικών στα πλαίσια καταναγκαστικών γάμων. Η Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης επίσης έχει εκδώσει ένα εγχειρίδιο ενημερωτικό όσον αφορά την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου. Όσον αφορά τώρα τις νύφες κατά παραγγελία και πώς αυτές τελικά μπορούν να μπλέξουν στα δίκτυα αυτά διακίνησης. Ήδη από το 2013 υπάρχει πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά την καταπολέμηση του φαινομένου αυτού στο διαδίκτυο. Κατά τη διάρκεια του 2016 θα υποβάλουμε συγκεκριμένες συστάσεις για το πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το διαδίκτυο ως όργανο πρόληψης και όχι ως όργανο στρατολόγησης των γυναικών αυτών. Τέλος, μαζί με τη Eurofound του Δουβλίνου εκπονούμε μια μελέτη για τον ρόλο των ε, υπηρεσιών ε, των γραφείων συνοικεσιών. Γιατί πολλές φορές έχουν γίνει καταγγελίες και για εργασιακή εκμετάλλευση των γυναικών αυτών. Περαιτέρω όμως αναλύσεις θα γίνουν προκειμένου να δούμε ποιες είναι οι βέλτιστες πρακτικές που υπάρχουν ήδη στα κράτη-μέλη και που θα, μπορούσαμε να μας, θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν να ρυθμίσουμε καλύτερα τη λειτουργία αυτή των γραφείων συνοικεσιών. Σε κάθε περίπτωση θέλουμε στα γραφεία αυτά, ακόμα και αν είναι νόμιμα, να καταπολεμήσουμε κάθε φαινόμενο εμπορίας ή εκμετάλλευσης των γυναικών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι πολύ σημαντικό επίσης να δούμε τι κάνουμε με τα κέρδη της εμπορίας ανθρώπων και να δούμε επίσης και ποια είναι τα επίπεδα προσφοράς και ζήτησης αυτής της ε, παράνομης ε, εμπορίας ανθρώπων. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε λοιπόν και τα παράνομα έσοδα τα οποία προκύπτουν. Ποιες θα είναι τώρα οι μελλοντικές μας εκθέσεις ε, όσον αφορά την διάσταση του φύλου στην εμπορία των ανθρώπων. Στα τέλη του 2015, τις αρχές του 2016, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει μια έκθεση όσον αφορά τη διάσταση του φύλου για την εμπορία των ανθρώπων. Επίσης θα παρουσιάσουμε την πρώτη μας έκθεση όσον αφορά την πρόοδο που έχει σημειωθεί για την καταπολέμηση εμπορία των ανθρώπων και το πώς η οδηγία έχει αρχίσει ήδη να εφαρμόζεται στα κράτη-μέλη. Μαζί με την έκθεση αυτή θα υποβάλουμε και άλλη μια έκθεση που θα έχει να κάνει με την ποινικοποίηση της εμπορίας ανθρώπων αν δηλαδή τα κράτη-μέλη έχουν επινικοποιήσει επαρκώς σχετικές υπηρεσίες ή όχι. Και επίσης προσβλέπουμε και στην οδηγία, έκθεση εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά την αντιμετώπιση της εμπορίας των ανθρώπων και θέλουμε επίσης να εκπονήσουμε και μια στρατηγική για μετά το 2016 όσον αφορά την αντιμετώπιση του φαινομένου της εμπορίας των ανθρώπων. Μέχρι τότε θα έχουμε τη δυνατότητα να λάβουμε υπόψη μας και τις παρατηρήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά και τις παρατηρήσεις και τη συμβολή των εθνικών κοινοβουλίων που νομίζουμε ότι θα πρέπει όντως να ενταχθούν ως αναπόσπαστα μέρη της νέας αυτής στρατηγικής για μετά το 2016. Στρατηγική για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων. Πρόεδρος, κοιτάξτε, πήρα στην αρχή το λόγο και θα μπορούσα και εγώ να πω κάποια πράγματα, αλλά ίσως να δώσω πρώτα το λόγο στην κυρία Ρένα σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ για όλες αυτές τις πληροφορίες. Το ζήτημα της οδηγίας για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων όντως μπορεί να είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο, πολύ χρήσιμο μέσο το οποίο πρέπει να αξιοποιήσουμε. Το ερώτημα όμως που θέσαμε στο παρελθόν ήταν το εξής. Αντί να λέμε ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη κάποιες υπηρεσίες, κάποιοι παράγοντες με ένα αμφίβολο ρόλο όσον αφορά την βιομηχανία αυτήν υφών κατά παραγγελία, είπαμε ότι θα έπρεπε να δούμε ποια εργαλεία εμείς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να σταματήσουμε πρακτικές ε, οι οποίες είναι πρακτικές διακινητών, παράνομες πρακτικές. Στην πράξη δηλαδή θέλαμε να δούμε πώς μπορούμε να αναλάβουμε δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να έχουμε καλύτερη ενημέρωση για τις γυναίκες και τις νέες κοπέλες που πέφτουν θύματα των δικτύων αυτών και δεύτερον να μπορούμε συγκεκριμένα να αναλάβουμε δράση κατά των γραφείων αυτών συνοικησιών. Να δούμε δηλαδή πώς μπορούμε να πλαισιώσουμε τη λειτουργία τους. Το ότι έχουμε κανόνες γενικά και αόριστα για την απασχόληση δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να πλαισιώσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα γραφεία αυτά. Αυτό ακριβώς κάνουμε γενικότερα και με την απασχόληση. Κάθε φορά που έχουμε γραφεία έβρεσης προσωρινής εργασίας προσπαθούμε να πλαισιώνουμε το ρόλο τους. Ε, θέλουμε και τώρα να πλαισιώσουμε το ρόλο των γραφείων αυτών συνοικεσιών τα οποία μπορεί σαφώς να λειτουργούν νόμιμα, αλλά θα πρέπει να ακολουθούν συγκεκριμένε νόμιμες πρακτικές και όχι εγκληματικές, παράνομες πρακτικές, όπως γίνεται πολύ συχνά. Και πολύ συχνά ξέρετε ότι θα πρέπει να κλείσουμε και κάποια τέτοια γραφεία, γιατί λειτουργούν εντελώ παράτυπα και εντελώ παράνομα. Ήθελα λοιπόν να πω ότι αυτά ήταν τα βασικότερα στοιχεία των ερωτημάτων που είχαμε απευθύνει προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Thank you. Um, I just want to add to that before I come to... Πρωτού περάσω σε άλλους ομιλητές, ήθελα να προσθέσω και εγώ κάτι. Η απάντησή σας εστιάζεται ε, στο θέμα της ε, παρατυπίας. Ε, όμως, πολλοί ε, γάμοι γίνονται μέσω του διαδικτύου ή μετά από διακοπές ε, και ε, είναι απολύτως νόμιμοι και κάποιοι επιτυχημένοι. Όμως, αυτό που μας ανησυχεί εμάς είναι ως πόσες έρχονται σαν ύφη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι απομονωμένοι, δεν γνωρίζουν τα δικαιώματά τους, δεν ξέρουν η Ευρωπαϊκή Ένωση τι τους προσφέρει. Δεν μιλάμε για λευκούς γάμους ή καταναγκαστικούς γάμους. Ξέρουμε ότι είναι παράνομοι και καλύπτονται από την νομοθεσία για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και ασχολούμαστε τώρα μάλιστα με την έκθεση υλοποίηση για την εμπορία ανθρώπων και θα κάνουμε πολλές συζητήσεις. Όμως δεν είναι αυτό που μας απασχολεί. Δεν, δεν ακούσαμε από εσάς κάτι σε σχέση με αυτή τη βιομηχανία νηφών μέσω διαδικτύου. Είναι παγκόσμιο ε, το φαινόμενο και έρχονται πολύ ευάλωτοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν φτιάξει σχέσεις ε, στο διαδίκτυο ή με επισκέψεις που έχουν κάνει, δεν τους υποχρεώνει κανείς και έρχονται ε, στην Ένωση χωρίς όμως να γνωρίζουν ποια νομοθεσία τους καλύπτει. Θα κάνετε μελέτη μας είπατε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε ποια είναι η κατάσταση και φυσικά ξέρουμε ότι υπάρχουν και διασυνδέσεις με τους εικονικούς γάμους και τους καταγκαστικούς γάμους και το παράνομο αυτό δίκτυο. Όμως μην ξεχνάτε και το νόμιμο κοπάτι, τους ευάλωτους ανθρώπους που δεν γνωρίζουν απλώς τα δικαιώματά τους. Είναι διαφορετικό, διαφορετική κατάσταση και διαφέρει από την εμπορία ανθρώπων και από τους ε, εικονικούς ε, γάμους. Η κυρία Μπελμπάου. Ευχαριστώ, Καθρίν. Και εγώ αυτή τη διάκριση ήθελα να κάνω, διότι βλέπουμε ότι δεν είναι ε, όλοι οι γάμοι ε, παράνομοι, αλλά για τους νόμους θέλουμε αρμονισμένα πρότυπα. Αυτό χρειαζόμαστε. Υπάρχει ένα κενό και αυτό πρέπει ακριβώς να καλυφθεί για να μην ε, ε, να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στην πραγματικότητα. Σε άλλες περιπτώσεις μπορούμε να προβλέψουμε τι θα συμβεί, αλλά όπως σωστά είπατε υπάρχουν ε, οι υπηρεσίες, πρακτορία που ασχολούνται με αυτήν την δραστηριότητα και θα έπρεπε να ξέρουμε με ποιο τρόπο θα μπορούσαμε να προστατεύσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω για την εφαρμογή της οδηγίας σε ποια είναι η κατάσταση στα 28 κράτη-μέλη. Διότι υπάρχουν οι οδηγίες αλλά δεν εφαρμόζονται ομοιόμορφα δεν υπάρχει παρακολούθηση, δεν υπάρχει αξιολόγηση. Οι πληροφορίες έχουμε αρκετές νομίζω, δεν μας χρειάζονται άλλε. Για να του θέλουμε να ασχοληθούμε με το ζήτημα της εμπορίας ανθρώπων. Είναι περίπλοκο το ζήτημα. Είναι σημαντικό λοιπόν να γνωρίζουμε την κατάσταση για να καταπολεμήσουμε αυτήν την απαράδεκτη συμπεριφορά. Χρειάζεται δίκαιη ανταλλαγή των ε, στοιχείων που έχουμε. ούτως ώστε να καταπολεμηθεί αυτό το φαινόμενο. Πηγαίνουν από χώρα σε χώρα αυτές οι γυναίκες ε, για να μην παραμείνουν υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα σε μία χώρα και ε, για να μην μπορέσουν να εντοπιστούν. Είναι ένα άλλο είδος εμπορίας ανθρώπων. Χρειαζόμαστε στοιχεία από τα κράτη-μέλη για αυτό το φαινόμενο. Τρίτον, πάλι σε σχέση με την ποινική διάσταση του ζητήματο και νομίζω ότι έχετε ασχοληθεί με την εξέταση αυτής της διάστασης, ε, μας μιλάτε για την πρόληψη κυρίως στο διαδίκτυο. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, για τους άντρες σκοπεύετε να κάνετε κάτι. Πρέπει να ρωτηθούμε τι συμβαίνει. Και διάβασα αυτή τη βδομάδα ε, κάτι απίστευτο. Στη Μούρσια στην Ισπανία ε, συνελήφθη μια ομάδα που ανάγκαζε ε, τις γυναίκες να εκπορνεύονται ε, γυναίκες που είχαν μικρά παιδιά που φύλαζαν ακόμη. και μπορούσαν αυτοί οι πελάτες που αγόραζαν αυτή την υπηρεσία να κάνουν ό,τι θέλουν με αυτές τις γυναίκες. Είναι ε, αδιανόητα βάρβαρο αυτό που συνέβαινε και θα ήθελα μέσω του ελέγχου να επιβάλλουμε την εφαρμογή των οδηγιών, να ανταλλάσσονται πληροφορίες Σήμερα μα απασχολεί η ανταλλαγή δεδομένων για την καταπολέμηση τρομοκρατία. Λοιπόν, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα δεδομένα για να καταπολεμήσουμε τα φαινόμενα πιο αποτελεσματικά. Θα ήθελα να ξέρω αν η Επιτροπή έχει στοιχεία στη διάθεσή τη και αν όχι να με τα στείλει γραπτό. Σα ευχαριστούμε και για να ακούσουμε τώρα τις απαντήσεις θα δώσουμε το λόγο στην κυρία Έσκετ, την εκπρόσωπο της Επιτροπής. Ευχαριστώ. Ξεκινώ με την τελευταία ερώτηση. Εφαρμογή τη οδηγία για το τράφικινγκ. Πρόκειται για νέα νομοθεσία, πολύ πρόσφατη. Η προθεσμία για την ενσωμάτωση έληξε το 2013. Μέχρι στιγμή έχουμε ενημερωθεί για την πλήρη μεταφορά από 27 μέλη Μόνο η Γερμανία μένει. Όσον αφορά τη μελέτη συμμόρφωσης ε, μετά από μεταφορά, θα έλεγα ότι μόλις τώρα ξεκινάει η εφαρμογή αυτή τη οδηγία στα κράτη-μέλη, γιατί πρόκειται, όπως είπα, για νέα οδηγία. Εμείς υπογραμμίζουμε ότι είναι καιρός ανάληψης δράσης. θέμα είναι τι θα κάνουμε μεταξύ άλλων για τη ζήτηση. Άρθρο 18 στην οδηγία τα κράτη-μέλη προσπαθούν να προλάβουν ακριβώς την, το εμπορίο ανθρώπων ε, στοχεύοντας την εξάλληψη της ζήτηση καταρχάς. Επίσης γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η πλειονότητα αυτών των νηφών είναι νόμιμη μιλάμε για νόμιμη μετανάστευση. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει εκμετάλλευση, ότι δεν υπάρχει βία ή ότι οι γυναίκες αυτές δεν θα γίνουν θύματα εμπορίου αφού μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειάζεται λοιπόν να εντοπίσουμε τα θύματα με την συνεργασία των οργανισμών για το άσυλο, των προξενείων κλπ. Πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή, μάλιστα, στη χορήγηση των θεωρήσεων. Τώρα, ο ρόλος των ενδιαμέσων πρόκειται για μια πολύ σημαντική οικονομική δραστηριότητα που έχει σχέση και με το εμπόριο ανθρώπων. Πρέπει να δούμε πώς θα μπορούσαμε ενδεχομένω να παρακολουθήσουμε και να, αλλά και να ρυθμίσουμε τη λειτουργία αυτών των εντό αγωγικών γραφείων συνοικισιών. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κύριε Πέρντερ, ευχαριστώ για την απαντήσή σα. Κοιτάξτε, το εμπόριο ανθρώπων το αντιμετωπίζουμε. Δεν είναι αυτό το πρόβλημά μα. Είναι θέμα μα, δηλαδή. Αυτό το οποίο θέλουμε από σας είναι να εξετάσετε τη νομική πτυχή. Δηλαδή, να φροντίσει η Κομισιόν, δηλαδή εάν πρέπει να νομοθετήσει προκειμένου η Κομισιόν, εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει, δηλαδή από κατά τα άλλα κάθε γάμος μπορεί να συνεπαγείται να συνοδεύεται με βία, διακρίσεις κλπ. Αυτά συμβαίνουν. Το θέμα είναι πώς γίνεται άνθρωποι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης να αποδέχονται να συνάψουν μακρόχρονη σχέση με κάποιον Ευρωπαίο. Εδώ πολλές φορές εμπλέκονται πολύ μεγάλα ποσά. Κάποιοι εξαπατώνται ενδεχομένω. Μπορεί να εξαπατώνται και οι αποδέκτες οι Ευρωπαίοι, αν θέλετε. Συνεπώς δεν μιλάμε εδώ για εμπόριο ανθρώπων, για τράφικινγκ. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Αν και μπορεί να είναι τα δύο θέματα αυτά συγκοινωνούντα δοχεία. Εμεί στη γραπτή ερώτηση μιλήσαμε για κάτι άλλο. Ρωτούσαμε την Κομισιόν τι κάνετε εσεί ω Κομισιόν σχετικά με τα δικαιώματα και τι ευθύνε των μεταναστών γυναικών που έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μπαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω αυτών των γραφείων και που μπορεί να μην γνωρίζουν δικαιώματα και υποχρεώσει και ευθύνε. Τι κάνετε λοιπόν επίση για να προστατεύσετε του Ευρωπαίου πολίτε τους οποίους κάποια γραφεία ενθαρρύνουν να αναζητήσουν ε, γυναίκες ή ζύγους μέσω αυτών των δικτύων. Επαναλαμβάνω δεν πρόκειται για τράφικινγκ, δεν είναι εμπόριο ανθρώπων. Παρά το γεγονός, επαναλαμβάνω, ότι μπορεί αυτά τα δύο να είναι σε ορισμένε περιπτώσεις συγκοινωνούντα δοχεία. Το αντιμετωπίζουμε λοιπόν ξεχωριστά. Χρειάζεται ή όχι νομοθέτηση εμπροκειμένου. Η μεσω αυτων των δικτυων επαναλαμβανω δεν προκειται για τραφικινγκ δεν ειναι εμποριο ανθρωπων παρα το γεγονος επαναλαμβανω οτι μπορει αυτα τα δυο να ειναι σε ορισμενε περιπτωσεις τα δοχεια το αντιμετωπιζουμε λοιπον ξεχωριστα χρειαζεται η οχι νομοθετηση εμπροκειμενου η κομισιον θα το δει λίγο πιο σοβαρά. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κύριε Μπέρτερ. Ζητώ από την Κομισιόν να απαντήσει στα σχόλια και τις ερωτήσεις και περνάμε στο επόμενο σημείο της μερικής διάταξης που είναι η έκθεση για την ισότητα των φίλων. η θέση των γυναικών στην ψηφιακή εποχή. παρακαλώ, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Όπως ξέρετε, είναι η δεύτερη φορά που συζητάμε το ζήτημα αυτό στην Επιτροπή μας. Κάναμε και μία δημόσια κρόση με τρεις ομιλητές. Νομίζω ότι ε, μας βοήθησε να καταλάβουμε τις διάφορες διαστάσεις του ζητήματος αυτού, η ακρόση που κάναμε και κατά την προετοιμασία της έκθεσης αυτής ήρθαμε σε επαφή με πολλές οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών που μας ενημέρωσαν για πολλές διαφορετικές πτυχές του ζητήματος αυτού. Νομίζω ότι έχουμε ήδη μια πάρα πολύ καλή βάση για να προχωρήσουμε λοιπόν και εμείς στη συζήτησή μας. Θα μπορούσα πολύ σύντομα να διατρέξω το κείμενο αυτό και να αφαιρθώ στα διάφορα ζητήματα που θέλουμε να αντιμετωπίσουμε στα πλαίσια αυτής της έκθεσης. Καταρχάς, ένα πολύ σημαντικό τμήμα της έκθεσης και μια βασική αρχή μας όπως βλέπετε και στον τίτλο, είναι να καταφέρουμε να ενδυναμώσουμε τις γυναίκες στην ψηφιακή εποχή. Το ζήτημα της ενδυνάμωσης λοιπόν είναι πολύ σημαντικό στοιχείο για μα. Θέλουμε να καταφέρουμε να δώσουμε περισσότερες ευκαιρίες και δυνατότητες στις γυναίκες στα πλαίσια μιας νέας ψηφιακής εποχής. Και οι γυναίκες με τη δικιά τους, από τη δικιά τους πλευρά μπορούν να συμβάλλουν σε αυτή τη νέα ψηφιακή εποχή. Θέλουμε λοιπόν να έχουμε μια επικοδομητική θετική προσέγγιση, αλλά παράλληλα λέμε ότι υπάρχουν και προβλήματα. Δεν πρόκειται να σας διαβάσω τώρα προφανώς την ε, έκθεση. Σας καλώ να το κάνετε εσείς, να δείτε την έκθεση αυτή γιατί έχει πολλά ενδιαφέροντα σημεία, να αναφερθώ τουλάχιστον στα πιο σύντομα, στα πιο σημαντικά σημεία. Καταρχάς, θέλουμε να δούμε πώς μπορούμε να ενσωματώσουμε την ισότητα των φύλων στην ψηφιακή ατζέντα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ξέρετε ότι το θεματολόγιο αυτό αποτελεί προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καταβάλλονται πολλές προσπάθειες, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν έχει επικεντρωθεί επαρκώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο ζήτημα της ισότητας των φύλων. Θέλουμε λοιπόν εμείς να δούμε πώς μπορούμε να ενσωματώσουμε τα ζητήματα των δικαιωμάτων των γυναικών και της ισότητας των φύλων στην ψηφιακή ατζέντα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είναι σε εξέλιξη. Προκειμένου λοιπόν να γίνει κάτι τέτοιο, διαρθρώσαμε την έκθεση αυτή, καταρχάς βάσει γενικών συστάσεων, Προσπαθούμε μέσω των γενικών αυτών συστάσεων να δώσουμε μια γενικότερη εικόνα του τι συμβαίνει και του πώς έχουν τα πράγματα και στη συνέχεια επικεντρωνόμαστε σε πιο εξειδικευμένα επιμέρου ζητήματα. Ασχολούμαστε με το ζήτημα της δημοκρατίας και της συμμετοχής στην ψηφιακή αυτή εποχή. Λέμε ότι αλλάζει η αγορά απασχόλησης, αλλάζει η εκπαίδευση, νέες ευκαιρίες κατάρτισης προκύπτουν και νέες οικονομικές ευκαιρίες. Και βέβαια έχουμε και κάποια προβλήματα, βία κατά των γυναικών ή άλλα αρνητικά φαινόμενα τα οποία υπάρχουν και στα πλαίσια της ψηφιακής εποχής. Όσον αφορά τη δημοκρατία και τη συμμετοχή, πιο συγκεκριμένα, θελήσαμε να επικεντρωθούμε στι πάρα πολλέ ευκαιρίε που προκύπτουν για μια ευρύτερη συμμετοχή των γυναικών μέσω νέων ψηφιακών μέσων και συγκεκριμένα προτείνουμε διαφορετικά εργαλεία τα οποία θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε, όπως για παράδειγμα το πρόγραμμα Ευρώπη για τους πολίτες ή ακόμα και κάποια άλλα εργαλεία ή κάποια άλλα μέσα. Καλό βέβαια και τους σκιώδεις συγητές να προτείνουν και νέα μέσα τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν προκειμένου οι γυναίκες να συμμετέχουν περισσότερο στην ψηφιακή εποχή. Επίσης ξέρετε ότι θα έχουμε και μια γνωμοδότηση από την Επιτροπή Απασχόλησης Ασχολούμεθα όμω και εμεί στην εκθεσή μα με το ζήτημα τη αγορά-εργασία. Έχουμε μια ψηφιοποίηση τη αγορά-εργασία που δεν επηρεάζει μόνο αυτού που εργάζονται στον τομέα τη πληροφορική, αλλά όλου του εργαζομένου σε όλου του κλάδου. Και υπάρχει βέβαια και μια ειδική διάσταση τη ισότητα των φύλων που πρέπει να ληφθεί υπόψη. Α μην ξεχνάμε ότι είναι οι γυναίκε αυτέ οι οποίε πλήττονται από τι επισφαλεί θέσει απασχόληση, από συμβάσει μερική απασχόληση, από εκτεταμένες ε, ώρες εργασίας ή από χαμηλές αποδοχές. Θέλουμε λοιπόν και αυτά τα στοιχεία να τα θίξουμε στην έκθεση και όταν βλέπουμε ότι 120.000 θέσεις απασχόλησης δημιουργούνται στον τομέα της πληροφορικής σε αιτήσια βάση, θέλουμε ορισμένες από τις θέσεις αυτές να απευθύνονται στις γυναίκες, έτσι ώστε οι γυναίκες να μπορούν να απασχολούνται περισσότερο σε αυτόν τον κλάδο. Περνάω στο επόμενο σημείο, εκπαίδευση και κατάρτιση. Πώς μπορούμε να δώσουμε ειδικά στις γυναίκες τις απαραίτητες δεξιότητες προκειμένου να λάβουν και αυτές μέρος ενεργά στην λεγόμενη ψηφιακή επανάσταση. Προσπαθούμε να δούμε τι κίνητρα μπορούμε να δώσουμε στις γυναίκες προκειμένου να ασχοληθούν με τα μαθηματικά και τις θετικές επιστήμες, πώς μπορούμε να προσεγγίσουμε εντελώ διαφορετικά το ζήτημα της πληροφορικής προκειμένου να καταρτίζονται στον κλάδο αυτό περισσότερες γυναίκες και προτείνουμε μάλιστα και ένα ευρωπαϊκό University Online στο διαδίκτυο έτσι ώστε όλο και περισσότερες γυναίκες από όλες τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης να μπορούν να καταρτίζονται σε ιδιαίτερα τεχνικά θέματα όπως αυτό της πληροφορικής. Θέλουμε από την άλλη να καταφέρουμε να ενσωματώσουμε όλο και περισσότερο ψηφιακές σπουδές ή ψηφιακά προγράμματα στα πιο συμβατικά εκπαιδευτικά προγράμματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν μιλάμε τώρα για επενδύσεις και επιχειρηματικότητα, η βιώσιμη ανάπτυξη, είναι πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι πάρα πολλά χρήματα δίνονται αυτή τη στιγμή στην ε, ψηφιακή ατζέντα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θέλουμε λοιπόν και εμείς από τη δική μα πλευρά να δούμε πώς μπορούν οι πόροι αυτοί να χρησιμοποιηθούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να προωθούν την ισότητα των φύλων. Αν έχουμε για παράδειγμα στοχευμένα ταμεία, στοχευμένου πόρους για τις γυναίκες επιχειρηματίες στον τομέα της πληροφορική, αυτό σίγουρα θα δώσει στις γυναίκες αυτές καταπληκτικές ευκαιρίες και θα οθήσει όμως και περισσότερες γυναίκες να συμμετέχουν στην ε, ψηφιακή αυτή τεχνολογία. Και τέλος, δεν θα πρέπει βέβαια να θελοτυφλούμε και μπροστά στα προβλήματα. Εξακολουθούμε και έχουμε πολύ σημαντικά προβλήματα βίας κατά, στο, κατά των γυναικών στο νέο αυτό ψηφιακό περιβάλλον. Λέμε λοιπόν στην έκθεση ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα φαινόμενα αυτά, αυτά τα προβλήματα, των οποίων τα, βαθικά, τα βαθύτερα αίτια πρέπει να ζητήσουμε στις ίδιες τις κοινωνίες μας, κυρίως στο αίσθημα μίσους κατά των γυναικών, στο γεγονός ότι ακολουθούμε ακόμα κάποια πατριαρχικά μοντέλα στις κοινωνίες μας. Πρέπει λοιπόν να καταφέρουμε να δείξουμε αλληλεγγύη προς τις γυναίκες, να υποστηρίξουμε τις γυναίκες για την καταπολέμηση αυτής της βίας. Προβλέπεται όμως και μια κατάρτιση αστυνομικών ή επαγγελματιών στο δικαστικό τομέα προκειμένου να γνωρίζουν καλύτερα πώς μπορεί να καταπολεμηθεί η βία κατά των γυναικών σε ένα ψηφιωμένο κόσμο, κυρίως όσον αφορά ορισμένες εφαρμογές στο διαδίκτυο. Ξέρετε ότι πολλές φορές έχουν γίνει καταγγελίες από γυναίκες και πολλέ φορέ οι ίδιοι αστυνομικοί, το δικαστικό προσωπικό που αντιμετωπίζει τι προσφυγέ αυτέ ή τι καταγγελίε, δεν γνωρίζουν καν τι είναι το Facebook ή πώ λειτουργεί το Facebook. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να υπάρχουν και τα απαραίτητα προγράμματα κατάρτιση αυτών των δημοσίων υπηρεσιών για να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε αυτά τα φαινόμενα βία. Έκανα μια πολύ σύντομη σφαιρική παρουσίαση τη κατάσταση. προσβλέπω στην συμβολή των ασκιωδών εισηγητών και ελπίζω ότι θα καταφέρετε να εμπλουτίσετε το σχέδιο αυτό έκθεση με περισσότερα σχόλια. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Μπιόρκ τώρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα της έκθεσης ε, και έλειπε αυτή η φεμινιστική σκόπια όταν εξετάζουμε το θέμα της ε, κοινωνίας ε, των ε, νέων τεχνολογιών. Είναι πάρα πολύ καλό, όπως λέει και η συγγύητρια, να διαπιστώσουμε με ποιο τρόπο μπορούμε να εξασφαλίσουμε νομοθεσία για ίση αμοιβή, λαμβάνοντα υπόψη όμω εξελίξει τη νέα αγορά εργασία με τι νέε τεχνολογίε. Ε, και μόνο έτσι μπορούν να έχουν επιρροή οι γυναίκε και να συμμετάσχουν στα δημοκρατικά δρόμενα. Όταν μιλάμε για εκδημοκρατισμό, ε, εγώ ακούω και ε, άλλα πράγματα. Παραδείγματο χάρη εκπαιδευτικά μέσα ανοιχτά. Μόνο έτσι μπορούμε να έχουμε μια δημοκρατική εκπαίδευση και καθολική πρόσβαση σε αυτά τα νέα μέσα και μπορεί να ασκήσει επιρροή η Επιτροπή μας ε, σε αυτό τον τομέα. Ε, θεωρώ δε ότι είναι περιεκτική η έκθεσή σας Ενδεχομένως ε, θα μπορούσαμε στο τμήμα συμμετοχή ε, και δημοκρατία να τονίσουμε και το ρόλο των ε, κοινωνικών μέσων δικτύωσης, των επιγραμμικών, δηλαδή Μπορούμε να διαρρήξουμε τα στερεότυπα και τον έλεγχο των αντρών στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και διαμόρφωση κοινή γνώμη, χρησιμοποιώντας ε, τις ψηφιακές πλατφόρμες και τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης. Αυτό μπορούμε να το ε, συζητήσουμε για τις απειλές ε, και για τα εγκλήματα, τα κύβερνα εγκλήματα είναι ξεκάθαρο, γιατί έχουμε ε, βιώματα στη Σουηδία, δηλαδή υφίστανται απειλές, οι γυναίκες ε, είναι πίσω από την οθόνη τους ε, και ξαφνικά νιώθουν ότι μπορεί από οποιαδήποτε στιγμή να δεχτούν απειλές. Οι αστυνομικές δυνάμεις όμως δεν αντιλαμβάνονται την κατάσταση δεν αντιλαμβάνονται ότι είναι πραγματικές οι απειλές που μπορεί να δεχτεί μια γυναίκα στο διαδίκτυο και ότι πρέπει να τις ερευνούν και να ακολουθούν τις συνέπειες συνήθει στις αστυνομικές διαδικασίες, όπως κάθε φορά που ε, δέχεται ε, σωματική απειλή, παραδείγματος χάρη μια γυναίκα. Θα συνεχίσουμε τις συζητήσεις για όλα αυτά τα ζητήματα ε, για να καταλήξουμε στι συναντικές λύσεις. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Αγιούτο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Στην έκθεση αυτή βλέπουμε πολλά θετικά στοιχεία πράγματα που μας βρίσκουν ε, σύμφωνος. Ξέρετε ότι στην Ιταλία πάρα πολλά πράγματα περνάνε από το διαδίκτυο. Βρισκόμαστε σε μια πολιτική φάση στην Ιταλία που βλέπουμε ότι μέσω του διαδικτύου μπορούμε τελικά να επηρεάσουμε πάρα πολύ την κατάσταση των ε, γυναικών. Πρέπει λοιπόν να εκμεταλλευτούμε θετικά τις ε, νέες αυτές ψηφιακές τεχνολογίες. Από την άλλη όμως, δεν θα πρέπει να θελοτυφλούμε μπροστά στους κινδύνους που μπορούν να προκύψουν μέσω του διαδικτύου. Κίνδυνοι βέβαια κυρίως για τις γυναίκες. Για παράδειγμα, πριν από λίγο καιρό στην Ιταλία είδαμε ότι υπήρχε ένας οργανισμός επιγραμμικός ο οποίος προσπαθούσε να προσιλητήσει μικρές ε, νέες γυναίκες για να τις εκμεταλλευτεί τελικά σεξουαλικά. Το διαδίκτυο με άλλα λόγια σου δίνει πάρα πολλές ευκαιρίες, διευρύνει τους ορίζοντες, αλλά παράλληλα σε καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτο. Και αυτό ισχύει πάρα πολύ για τις νέες γυναίκες, για τα κορίτσια, για τις κοπέλες. Αν λοιπόν δεν υπάρχει απαραίτητη επιτήρηση, απαραίτητη παρακολούθηση, αν δεν υπάρχει απαραίτητη υποστέριξη από τις ίδιες οικογένειες, Πολύ συχνά μιλάμε βέβαια για κορίτσια τα οποία είναι μόνα τους μπροστά στην οθόνη. Αν δεν υπάρχει πλαισίωση αυτή, τότε ελοχεύει ο κίνδυνος να αποτελέσουν οι γυναίκες αυτές θύματα εκμετάλλευσης. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν, όπως είπατε, να υπάρχει απαραίτητη κατάρτιση όσον αφορά τον ψηφιακό αυτό κόσμο. Πολύ συχνά υπάρχει ένα χάσμα πλέον μεταξύ γονέων και παιδιών οι γονείς δεν γνωρίζουν πολλές φορές τις ευκαιρίες αλλά και τους κινδύνους που κρύβουν οι νέες τεχνολογίες. Τα παιδιά μας, η νέα αυτή γενιά του iPad, δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί, πώς θα είναι μετά από 20 χρόνια. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει ήδη από τώρα να καταφέρουμε να ενημερωθούμε καταλήλως και να βοηθήσουμε να δώσουμε προς τους νέους τις απαραίτητες πληροφορίες, την καλύτερη δυνατή ενημέρωση όσον αφορά την ψηφιακή αυτή εποχή. Είναι πολύ σημαντικό να διευκολύνουμε την πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες, αλλά αυτή να πρέπει να είναι προστατευόμενη. Από την άλλη έχουμε 20 εκατομμύρια ακόμα Ιταλών οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση καν στο διαδίκτυο. Ας μην ξεχνάμε λοιπόν ότι υπάρχουν ακόμα πάρα πολλοί πολίτες οι οποίοι όχι μόνο δεν χρησιμοποιούν το διαδίκτυο, αλλά δεν έχουν στοιχειώδη ενημέρωση όσον αφορά τις διαφορετικές πτυχές του. Πρέπει λοιπόν να προωθήσουμε και έναν γραμματισμό ψηφιακό. Θεωρώ ότι το σχέδιο αυτό έκθεσης είναι πολύ θετικό και εμείς θα το υποστηρίξουμε. Θεωρούμε ότι έχετε δημιουργήσει ήδη μια πολύ θετική πρώτη βάση. Ευχαριστώ. Eh. Ευχαριστούμε πολύ παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω την εισηγήτρια. Προφανώς εργάστηκε πολύ καλά για την έκθεση αυτή, φαίνεται αυτό, και είχαμε και μια πολύ ευρεία συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους. Θεωρώ λοιπόν ότι καταλήξαμε σε μια έκθεση η οποία είναι πολύ καλά διαρθρωμένη και περιέχει πολύ θετικά στοιχεία. Πιο συγκεκριμένα, γίνεται πολύ σωστά αναφορά στην έκθεση αυτή σε διάφορες πτυχές που έχουν να κάνουν με τις ευκαιρίες καταρχάς που έχουν οι γυναίκες στη νέα ψηφιακή εποχή. Ευκαιρίες προκύπτουν από το νέο αυτό ψηφιακό περιβάλλον. Πολύ σωστά έκανε και τις εντόπισε τις ευκαιρίες αυτές η συγγήτρια. Επίσης, πολύ σωστά εντόπισε όμως και τις απειλές και τους κινδύνους που πλήττουν τις γυναίκες, όπως η βία στο διαδίκτυο. Θα ήθελα παρόλα αυτά να κάνω και εγώ κάποιες περαιτέρω παρατηρήσεις. Πέρα λοιπόν από τα αρχικά αυτά συγχαρητήρια, να σας ευχαριστήσω για την μνήα που κάνετε στις υφιστάμενες εκθέσεις και τις υπάρχουσες δηλώσεις όσον αφορά το ζήτημα αυτό. Όσον αφορά τα πιο αφιλεγόμενα ζητήματα τώρα, δεν συμφωνώ πλήρως με την αξιολόγηση που κάνετε όσον αφορά τους κινδύνους, κίνδυνοι στις οποίες, στους οποίους εκτίθενται οι γυναίκες, ιδίως στα πλαίσια του διαδικτύου. Αναφερθήκατε εδώ πέρα σε επισφαλείς θέσεις απασχόλησης, σε θέσεις απασχόλησης με χαμηλές αποδοχές. Πού βασίζεστε ακριβώς για να κάνετε τέτοιες δηλώσεις, γιατί η έρευνα που έχουμε από άλλες εκθέσεις, ή μελέτες, μας δείχνουν ότι τα πράγματα είναι διαφορετικά. Η συγγήτρια επίσης αναφέρθηκε στις αρνητικές επιπτώσεις στην εξισορρόπηση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής εξαιτίας της ψηφιακής εποχής. Με εμπειρία μου μου δείχνει ακριβώς το αντίθετο. Η ψηφιακή εποχή μας επιτρέπει την τηλεεργασία, τις πιο ευέλικτες μορφές εργασίας, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι διευκολύνονται οι γυναίκες και οι άντρες να εξισορροπήσουν προσωπική και επαγγελματική ζωή. Πάλι λοιπόν ζητάω από την εισηγήτρια να μου δώσει κάποιες διευκρινήσεις. Ποιες είναι οι πηγές σας. Πώς μπορείτε να λέτε ότι η ψηφιακή εποχή δεν βοηθά τη συμφιλίωση προσωπικής επαγγελματικής ζωής. Θα υποβάλουμε εκ μέρους του ΕΛΚ επίσης και κάποιες α, περαιτέρω τροπολογίες. Ιδίως όσον αφορά το ζήτημα της επικουρικότητας. Σε πάρα πολλά σημεία αναφέρεστε σε αρμοδιότητες οι οποίες είναι καθαρά εθνικές. Ας είμαστε λοιπόν πάρα πολύ προσεκτικοί και ας την αρχή της επικουρικότητας. Όσον αφορά τώρα τα ζητήματα αυτά τα οποία θα πρέπει να αναπτύξουμε και να βελτιώσουμε στα πλαίσια της έκθεσης. Πρώτο, εντοπισμός νέων ευκαιριών. Ευκαιρίες που έχουν να κάνουν με την ψηφιοποίηση των χωρών μας. Νέες δυνατότητες προκειμένου να δυναμωθεί ο ρόλος των γυναικών στην ψηφιακή εποχή. Ας μην ξεχνάμε ότι ε, ο ψηφιακό κλάδος συνήθως έχει θέσει απασχόληση, οι οποίες πληρώνονται πολύ καλά. Κατά αυτόν τον τρόπο, εφόσον οι γυναίκε εργάζονται στον κλάδο αυτό, θα μπορέσουν να μειώσουν και το χάσμα το μισθολογικό που τις χωρίζει με τους άντρε. Όσον αφορά τώρα την επιχειρηματικότητα των γυναικών, αυτό το οποίο δεν μου αρέσει εδώ πέρα είναι ότι αναφέρεστε εσείς σε μια ξεχωριστή ακαδημία που θα πρέπει να δημιουργηθεί προκειμένου να αυξηθεί ο γραμματισμός των γυναικών, όπως λέτε. Λίγο ατυχές είναι αυτό. Μήπως θα έπρεπε να λέτε καλύτερα ότι θα πρέπει να δοθούν ε, επιδοτήσεις στις γυναίκες, χρηματοδότηση, υποτροφίες προκειμένου να καταφέρουν να αυξήσουν ε, τις ψηφιακές τους δεξιότητες όσον αφορά επίση την επιχειρηματικότητα των γυναικών. Μήπω θα έπρεπε να αναφερθείτε εδώ πέρα και στην κοινωνική οικονομία, γιατί και στα πλαίσια τη οικονομία αυτή θα δημιουργούνταν νέε ευκαιρίε για τι γυναίκε να ανοίξουν κάποιε νέε επιχειρήσει. Και όσον αφορά τώρα την ε, βία και τη διάσταση των φύλων, Ξέρετε ότι έχουμε και τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, την οποία δεν αναφέρεται και η οποία όμως ε, περιλαμβάνει κάποια πολύ θετικά επιχειρήματα τα οποία θα στήριζαν τα όσα λέτε εσείς στην έκθεσή σας. Να αναφερθώ επίσης και στην ε, βία αυτή κατά των γυναικών, καθώς επίσης και στην σεξουαλική εκμετάλλευση των ε, κοριτσιών. Τα όσα συμβαίνουν σε διάφορες χώρες είναι πραγματικά αποτρόπαια, η βλέπουμε ότι το διαδίκτυο πάρα πολλές φορές προωθεί στην κυρολεξία την εκπόρνευση των ε, νέων κοριτσιών. Πρόκειται για δίκτυα τα οποία είναι όλο και πιο διαθέσιμα, εντελώς ανώνυμα και βλέπουμε ότι υπάρχουν ε, πολλοί έφηβοι, παιδιά ή και φοιτητές που χρησιμοποιούν τέτοια δίκτυα ή που πέφτουν θύματα τέτοιων πρακτικών. Προφανώς δεν λέω ότι θα πρέπει να καταργήσουμε το διαδίκτυο, αλλά χρειαζόμαστε μια συνετή χρησιμοποίηση του διαδικτύου όπου θα προστατεύονται οι πιο ευάλωτες ομάδες όπως τα παιδιά. Υπάρχουν κάποια πολύ ύποπτε sites, ύποπτε ιστοσελίδες, στα πλαίσια των οποίων μπορούν κάποια παιδιά, νέοι ακόμα, να ανεβάζουν γυμνές φωτογραφίες. Ας είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, ας προσπαθήσουμε να ρυθμίσουμε αυτή τη χρήση του διαδικτύου. Να αναφερθώ τώρα επίσης και σε κάποια επιμέρους σημεία της έκθεσης αυτής, σε κάποια άρθρα σας. όπου κάνετε αναφορά πρώτον στο ζήτημα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. αφιερώνεται εσείς ένα ολόκληρο κεφάλαιο στην εκθεσή σας. Νομίζω ότι θα πρέπει να αφαιρθούμε περισσότερο στο ρόλο των καθηγητών και των δασκάλων. Η διαπαιδαγώγηση δεν είναι πανάκια. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε υποστήριξη και για τους ίδιους τους καθηγητές. Χωρίς τους καθηγητές δεν πρόκειται να δούμε κανένα θετικό αποτέλεσμα στα σχολεία μας. Υποστήριξη λοιπόν όχι μόνο για τους μαθητές, υποστήριξη και για τους διδάσκοντες. Σας ευχαριστώ επίσης για τα όσα είπατε για την χρηματοδότηση της ε, επιχειρηματικότητας, ιδίως των ε, γυναικών επιχειρηματιών. Πρέπει όντως να τονίσουμε περισσότερο ότι υπάρχει ανάγκη για αυτή τη χρηματοδότηση. Στο άρθρο 20 αναφέρεστε σε κάποιους νέους πόρους που θα μπορούσαν να δοθούν για την ε, πρόθεση επιχειρήσεων που απασχολούν γυναίκες ή που δημιουργούνται από γυναίκες. Δεν νομίζω ότι από νομικής πλευράς θα ήταν δυνατόν κάτι τέτοιο όμως σε καμία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήμουν λοιπόν εγώ περισσότερο προσωπική με τέτοιες προτάσεις. Αυτά είχα να πω. Πέρα από όλα αυτά βέβαια πρέπει να πω ότι η έκθεσή σας είναι ιδιαίτερα πλήρης, κάνει πάρα πολλές προτάσεις και επίσης προχωρά σε μια πολύ σωστή διάγνωση της όλης κατάστασης. Να σε ευχαριστήσω λοιπόν για άλλη μια φορά για την έκθεσή σας αυτήν. Ευχαριστώ. Να είμαι σύντομη διότι τα σημαντικότερα ήδη ακούστηκαν. Λοιπόν, συγχαρητήρια στην κυρία και για την ε, εισηγησή της. Η ακρόαση ήταν πολύ ενδιαφέρουσα το του θέματος. Οι ομιλητές είπαν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, μίλησαν για νέα εργαλεία, κατέθεσαν καινοτόμες ιδέες, συνεισέφεραν στην έκθεση, το είπε άλλωστε και η συγγήτρια. Συνεπώς, δεν υπάρχει λόγος να παραλάβουμε τα γνωστά, σύμφωνα με τις περισσότερες απόψεις. Ε, σε Δύο θέματα μόνο να δύο λόγια, κυρία Μίλησε για το διαδίκτυο και τα παιδιά. Εγώ θα ήθελα αυτά να τα συνδέσω με την βία που έχει με το φύλλο. Διότι έχουμε στοιχεία, ξέρετε, αυτήν την νέα πραγματικότητα στην οποία οι νέοι επαναλαμβάνουν συμπεριφορές που υπό κανονικές συνθήκες δεν θα θεωρούσαν αποδεκτές. Δηλαδή μεταχειρίζονται τα νερά κορίτσια ως αντικείμενα, αν θέλετε. Και αυτά τα προάγει το διαδίκτυο. Αυτές οι συμπεριφορές διαδίδονται μέσω του διαδικτύου και αυτό είναι το πρόβλημα, ότι οι νέοι άνθρωποι απορροφούν, τέλος πάντων γίνονται κοινωνία αυτών των πρακτικών. Δεν ξέρω αν εδώ μπορούμε να προτείνουμε μια στρατηγική πρόληψης ή να δρομολογήσουμε μια εκστρατεία για να σταματήσουμε αυτή την ιστορία. Πιστεύω ότι είναι πραγματικά ανησυχητικό. Τι μπορούμε να κάνουμε όμως. Πρόκειται για θέμα συμπεριφοράς των νέων ανθρώπων που προάγονται μέσω διαδικτύου και που κατατείνουν σε βία βαρας των γυναικών. Η έκθεση, εν πάση περιπτώσει, είναι μια ευκαιρία θα βοηθήσει τις γυναίκες στην ψηφιακή εποχή. Να τονίσουμε επίσης την πτυχή της κατάρτισης, ιδιαίτερα σε συγκεκριμένους τομείς, ώστε οι γυναίκε να έχουν στα χέρια του περισσότερε ευκαιρίε στι αγροτικέ περιοχέ μάλιστα, είναι εξίσου σημαντικό να έχουν πρόσβαση σε νέε τεχνολογίε μέσω διαδικτύου. Η πρόσβαση αυτή δεν είναι παντού εγγυημένη βεβαίω, Εξού και το πρόβλημα. Η κατάρτιση πάντω θα ωφελήσει, αυτό είναι σίγουρο. Α δώσουμε ευκαιρίε, σε περισσότερε γυναίκε, α πούμε τηλεεργασίας. Έτσι όλες οι γυναίκες θα υποφεληθούν από τις νέες τεχνολογίες και το διαδίκτυο. Μην ξεχνούμε επίσης τις γυναίκες με αναπηρίες. Κάθε φορά που καταρτίζουμε προγράμματα, σαν τα προγράμματα στο πλαίσιο του Ταμείου Συνεχής, υπάρχουν εκπαιδεύσεις, καταρτήσεις για ευάλωτες ομάδες. Να σε αξιοποιήσουμε λοιπόν αυτά τα πρόγραμματα στο μέγιστο υπέρ των γυναικών με αναπηρίες, έτσι ώστε να υποφεληθούν και αυτές από τις τρέχουσες ευκαιρίες και να γίνουν ανταγωνιστικέ στην αγορά εργασία. Αυτά ήθελα απλώ να πω, λέει ο πρόεδρος. Και τώρα ο λόγος και πάλι στην εισηγήτρια για να σχολιάσει και να απαντήσει. Ευχαριστώ πρόεδρε, ευχαριστώ τους σκιώδει που έλαβαν τον λόγο. Πάρα πολλά από αυτά που είπατε ευχαρίστως να τα περιλάβουμε στην έκθεση. Να απαντήσω όμως ε, σε μερικές ερωτήσεις και να δώσω και μερικές διευκρινήσεις. Το πρώτο είναι αυτό που είπατε. Οι αρνητικές επιπτώσεις της ψηφιοποίησης της αγοράς, της αγοράς εργασίας. Υπάρχει μελέτη συνδικάτου η οποία δείχνει ότι η συμμετοχή στον χώρο εργασίας λόγω ψηφιοποίησης λόγω του διαδικτύου αντιμετωπίζει προβλήματα. Είναι και αυτό μια εξέλιξη που πρέπει να μα απασχολήσει. Όσον αφορά τα επιγραμμικά, τα διαδικτυακά πανεπιστήμια, Προφανώ δεν είναι μόνο για γυναίκε, είναι, είναι ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, τα οποία μπορούμε να αξιοποιήσουμε μαζί με διαδικτυακά εργαλεία, ακριβώς να παράσουμε εκπαίδευση και κατάρτιση, αλλά και να δώσουμε υποτροφίε σε γυναίκε. μπορούμε να συμπεριλάβουμε και άλλα σχόλια. Για την χρηματοδότηση πιστεύω ότι πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να παρέχουμε κίνητρα. Δηλαδή να εξασφαλίζουμε χρηματοδότηση σε γυναίκες, σε γυναίκες επιχειρηματίας μέσω στοχευμένων προγραμμάτων. Τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία και το κοινωνικό και το περιφερειακής ανάπτυξης έχουν αναπτύξει σχετικά εργαλεία και μπορούν να χρηματοδοτήσουν. Φυσικά στις μέρες μας συνεχίζουμε να παρατηρούμε ότι η συντριπτική πληρότητα των κονδυλίων πηγαίνει σε άντρε. Και όμω οι γυναίκε έχουν ιδέες, θέλουν να προχωρήσουν, να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Αυτά μπορούμε να τα συζητήσουμε ε, με την ευκαιρία της ζήτησης για το άρθρο 20 στη συνάντηση των σκιωδών. Ευχαριστώ για τα σχόλια και προσβλέπω σε μια επικοδομητική συζήτηση. Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ για να κλείσουμε με αυτό. σα ε, ενημερώνω για το χρονοδιάγραμμα. 16 Δεκεμβρίου υποβολή τροπολογιών. 17 Φεβρουαρίου ψηφίζουμε στην Επιτροπή. 17 Φεβρουαρίου και στην Ολομέλεια θα πάμε τον Απρίλιο του 2016. Αυτά λοιπόν. Κλείνει έτσι η πρωινή συνεδρία. Σα ευχαριστώ πολύ. Και συνεχίζουμε με τους συντονιστές. Παρακαλώ οι συντονιστές να μην φύγουν. Και παρακαλώ τους άλλους να φύγουν για να ξεκινήσει αμέσως η επόμενη συνεδρία. Ευχαριστώ.